Goedemiddag collega's. Eh, welkom allemaal. Καλώς ορίσατε όλοι σα στην ε, συνεδρίαση του ελέγχου του προπολογισμού που θα διαρκήσει δύο ημέρες, σήμερα και αύριο. Θα συνεδρια... Εγώ θα προεδρεύσω σήμερα το απόγευμα γιατί ο κύριος Δεμαντζίστρης θα έρθει αύριο. Έχουμε ένα σωρό ψηφοφορίες και ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα γίνουν ε, με χαρά και κέφι. Πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Υποθέτω ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες, δεν υπάρχουν ε, αλλαγές. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια σας παρακαλώ ετοιμάστε τις κάρτες ψηφοφορίας. διότι στην τελική ψηφοφορία της κάθε έκθεσης θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Όπως ξέρετε η συνεδρίαση αναμεταδίδεται απευθείας. Να είστε όλοι και σας και όλες σας ευγενικοί, διότι μας ακούνε και παρά έξω. Και στο σημείο 3 έχετε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας. της 10ης Φεβρουαρίου και τα λάβατε όλα αυτά στις 14 Μαρτίου. Λοιπόν, άμα δεν έχετε παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, εγκρίνονται τα πρακτικά. Πάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης σειράς ψηφοφοριών εκθέσεων του κυρίου Σταυρακάκη. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Σταυρακάκη πριν από την ψηφοφορία, όχι. Okay. dan gaan we naar het Πρώτη έκθεση. Στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Μεταφραστικό κέντρο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Πρόταση απαλλαγής υπέρ. Κατά. Α, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 12 υπέρ, 2 κατά και μία αποχή εγκρίνεται. Στη συνέχεια Εκαθάριση λογαριασμών. Πάλι ηλεκτρονικά ή πέρα κατά αποχές, πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα το ίδιο πράγμα. 12-2-1. Το ψήφισμα πάλι ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας 13.1.2 εγκρίνεται σημείο 5 Σεντεφόπ πάντα ηλεκτρονικά πρόταση απαλλαγής πάντα ηλεκτρονικά γιατί πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τα αποτελέσματα Πέρας ψηφοφορίας. 13-1-2. Εγκρίνεται. Πρόταση απόφασης. Υπέρ. Συγγνώμη, ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 14-1-1. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια έχετε τρεις τροπολογίες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι οι τροπολογίες 3 και 5 οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί ήδη στην έκθεση στα βρακάκι. Οπότε μένουν να ψηφίσουμε οι τροπολογίες 1, 2 και 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία του ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, ένας κατά και μία αποχή. Σημείο 6. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου της Αλίας. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για την πρόταση απαλλαγής. Η, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, κανένας κατά και δύο αποχές. Εκαθάριση λογαριασμών, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ και μία αποχή. Το ψήφισμα Έχουμε μία τροπολογία της Επιτροπής Αλίας, τροπολογία 3. Οι 1, 2 και 4 έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην έκθεση. Διάτανα των χειρών. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 17 υπέρ ένας κατά. Ε, ένας αποχή, συγγνώμη. Σημείο 7. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Μεταφορών. Έχουν ληφθεί υπόψη ήδη οι τροπολογίες. Πρόταση για την απαλλαγή αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ 2 αποχές. Καθάρις λογαριασμών ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 16 υπέρ. Κανένας κατά και μία αποχή. Τέσσερις τροπολογίες της Επιτροπής Μεταφορών. Θα ψηφίσουμε unblock. Άρση της χειρός κατά αποχές εγκρίνονται τελική ψηφοφορία του ψηφίσματος ηλεκτρονικά αρχίζει πέρας της ψηφοφορίας 17 υπέρ κανένας κατά και μία αποχή σημείο 8 Τροπολογία της 3, 4 και 10 της Επιτροπής Περιβάλλοντος έχουν συμπεριληφθεί. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την πρόταση απαλλαγής υπέρ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 16 υπέρ, κανένας κατά και δύο αποχές. Ε, καθάριση λογαριασμών, ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 1 κατά καμία αποχή. Έχουμε 7 τροπολογίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος Αμπλοκ Διαντάσεως της Χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, 18 ψηφίσαντες, μία αποχή. Σημείο 9. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων. 1, 2 και 7 της Επιτροπής Περιβάλλοντος έχουν συμπεριληφθεί. Πρέπει να ψηφίσουμε τις 4, 5 και 6, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε καταρχήν την απαλλαγή. Αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, κανένας εναντίον και δύο αποχές. Καθάριση λογαριασμών, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας 18 υπέρ και κανείς εναντίον καμία αποχή. 3, 4, 5, 6 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αμπλοκ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται ομόφωνα. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας 17 υπέρ, κανένα εναντίον, μία αποχή. Σημείο 10. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Έχουμε τροπολογίες Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η 4 έχει συμπεριληφθεί στο κείμενο, ένα κομμάτι της τροπολογίας 6 και τροπολογία 9. Σε λίγο δηλαδή θα πρέπει να ψηφίσουμε ορισμένε τροπολογίες. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά την απαλλαγή υπέρ. Ή μάλλον καλύτερα αρχίζει η ψηφοφορία, διορθώνει το πρόεδρο. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ, δύο αποχές, Κανένα εναντίον. Πρόταση για την εκαθάριση των λογαριασμών, το κλείσιμο μάλλον των λογαριασμών, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, μία αποχή. Οι τροπολογίες σαν Υπάρχει μία μικροαλλαγή, αλλά καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Είναι στο σημείο 6. Όλες τις τροπολογίες θα τις ψηφίσουμε αμπλόκ δεν βλέπω αχυρίς διανατάσσω στις χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ομόφωνα. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 20 ψηφίσανε υπέρ και μία αποχή. Καμία ψήφος κατά. Όλα βαίνουν καλώς. Σημείο 11. η Λίμπε έχει παρουσιάσει μια τροπολογία η οποία έχει συμπεριληφθεί στο κείμενο απαλλαγή λοιπόν ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας 17 υπέρ μία ψήφος κατά και δύο εποχές εγκρίνεται κλείσιμο λογαριασμών πάντα ηλεκτρονικά αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 19 υπέρ ένας κατά μία εποχή Έχουμε τρεις τροπολογίες της ΛΥΜΠΕ, ένα, τέσσερα και τρία. Μπορώ να τις περάσω αν μπλοκ διανατάσεως της χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 18 ψήφισαν υπέρ, ένας κατά και μία αποχή. Σημείο 12. Η ασφάλεια στη θάλασσα. 3, 4, 5, 6, 7, 8 της Επιτροπής Μεταφορών ήδη έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο. Ψηφίζουμε την πρόταση απαλλαγής, ηλεκτρονικά αρχής ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, 19 υπέρ, κανένας κατά και δύο αποχές το κλείσιμο των λογαριασμών ηλεκτρονικά αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 19 υπέρ μία αποχή δύο τροπολογίες της Επιτροπής Μεταφορών ένα και δύο τις ψηφίζουμε αμπόκ διανατάσεως της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, μία ψήφος κατά. Σημείο 13. Η ενίσα. Ηλεκτρονικά. Πρόταση απαλλαγή. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία 17 υπέρ, Ένα κατά δύο αποχές κλείσιμο των λογαριασμών, ηλεκτρονικά αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Ο κύριος Φέλνερ Αρίβ, αργήσατε κύριε Φέλνερ. 19 υπέρ, ένας κατά μία αποχή. Ο κύριος Φέλνερ θα συμμετέχει στη ψηφοφορία για το ψήφισμα, αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, ένας κατά μία αποχή. Σημείο 14. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, η ΕΡΑ. Έχουμε τις τροπολογίες 1, 3, 5, 6, 7, 8 και 9 που έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο. Είναι τροπολογίες Επιτροπής Μεταφορών και έχουμε λίγες τροπολογίες για μετά. Ψηφίζουμε για την απαλλαγή ηλεκτρονικά, αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 2 αποχές, κανένας κατά. Το κλείσιμο των λογαριασμών, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ και μία αποχή. Στη συνέχεια έχουμε μία τροπολογία, τις δύο, δύο καλύτερα, είναι οι δύο τροπολογίες Επιτροπής Μεταφορών διανατάσσεως της χειρός ψηφίζουμε μπλοκ. Κατά αποχές. Άμα λάθος έκανα λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη θα ψηφίσουμε πρώτα την δύο υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1 είναι η προφορική τροπολογία Κορνέλης Δε και ο εισηγητής συμφωνεί με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Έχω αμφιβολίες. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Για την παράγραφο 1. Αποτέλεσμα 9 υπέρ 12 κατά καμία αποχή απορρίπτεται. Στη συνέχεια η τροπολογία 4 της Επιτροπής Μεταφορών διανατάσσεως της χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, κανένας κατά και δύο αποχές. Σημείο 15. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή Απασχόλησης έχει καταθέσει δύο τροπολογίες, τη δύο και τη τρία έχουν συμπεριληφθεί και έχουμε να ψηφίσουμε άλλες δύο τροπολογίες μετά. Απαλλαγή καταρχήν. Ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, ένας κατά δύο αποχές. Ηλεκτρονικά το κλείσιμο των λογαριασμών αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας 19 υπέρ 1-1 το σκορ. Τροπολογίες της Επιτροπής Απασχόλησης Αμπλοκ για να τάσω στις χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, ένας κατά μία αποχή εγκρίνεται. 16. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία τροπολογίες τη Επιτροπής Απασχόλησης, τις έχουμε ήδη στο κείμενο 1, 2, 3 και 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 19 υπέρ, ένας κατά μία αποχή. Κλείσιμο λοιπόν των λογαριασμών, ηλεκτρονικός έλεγχος. ψηφοφορία ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 1 κατά, μία αποχή. Έχουμε μια τεχνική τροπολογία γιατί η τροπολογία 3 δεν χρειάζεται να τεθεί σε ψηφοφορία και φτάνουμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Με την κάρτα σας παρακαλώ ψηφίζουμε. Τέλος. 19 υπέρ, 1 κατά μία αποχή. Στο σημείο 17 τώρα. Έχουν ήδη γίνει δεκτές οι τροπολογίες της ε, Επιτροπής Απασχόλησης. Θα έχουμε άλλες δύο να ψηφίσουμε μετά. Θα θέσουμε σε ψηφοφορία την απαλλαγή πρώτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 20 υπέρ, ένας κατά, δύο αποχές. Στη συνέχεια ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κρίσιμο υπέρ. 21 ε, υπέρ, 1 κατά μία αποχή. Σχέδιο ψηφίσματος. Έχω δύο τροπολογίες Επιτροπής Απασχόλησης, την 3 και την 4. Μπορώ να τις ψηφίσουμε μαζί. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Τελική ψήφος τώρα. Τέλος. 20 υπέρ, 1 κατά, μία αποχή. Στο σημείο 18 τώρα φτάνουμε για το Eurojust. Δύο τροπολογίες της ΛΥΜΠΕ θα τις ψηφίσουμε μετά. Πρώτα θα ψηφίσουμε την πρόταση απαλλαγής. Τέλος. 21 υπέρ, 1 κατά μία αποχή. Δεύτερη ψηφοφορία. Τέλος. 21 υπέρ, 1 κατά. Καμία αποχή αυτή τη φορά. Τώρα οι δύο τροπολογίες της ΛΥΜΠΕ, οι 2 και οι 5, μαζί ψηφίζουμε παρακαλώ ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και οι δύο γίνονται δεκτές. Τελική ψήφος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 22 υπέρ, 1 κατά, καμία εποχή. Τώρα στο 19 για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει καταθέσει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τρεις τροπολογίες, η 1, 2 και 3 είναι ήδη στο κείμενο. Θα θέσουμε πρώτα σε ψηφοφορία την πρόταση απαλλαγής. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, 19 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Τώρα για το κλείσιμο των λογαριασμών. Τέλος. 20 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Το σχέδιο ψηφίσματος τώρα μας οδηγεί στην ψηφοφορία της 4 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα παράγραφος 4 με προφορική τροπολογία De Jong. Ο εισηγητής συμφωνεί με την τροπολογία αυτή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τελική ψήφος με την κάρτα. Τέλος. 20 υπέρ, 3 κατά. Περνάμε τώρα στο σημείο 20. για το GNSS. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι σημαίνει GNSS, αλλά έτσι το λέμε όλοι, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζουμε κάτι ο καθένας. Θα ψηφίσουμε τώρα για την απαλλαγή. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 20 υπέρ, 1 κατά δύο αποχές. Τώρα για το κλείσιμο των λογαριασμών του GNSS ψηφίζουμε. Τέλος, 20 υπέρ, ένας κατά μία αποχή. Τώρα στο σχέδιο ψηφίσματος έχω δύο τροπολογίες προφορικές. De Jong. Ο εισηγητής συμφωνεί με τις προφορικές αυτές τροπολογίες, τις ψηφίζουμε μαζί. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, οι τροπολογίες γίνονται δεκτές. Τελική ψήφος με την κάρτα. Τέλος. 20 υπέρ, ένα κατά, μία αποχή. Στη συνέχεια περνάμε στο σημείο 21 για το Artemis. Κοινή δράση. Πρόταση απαλλαγής, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 19 υπέρ, ένας κατά, δύο απέχουν. Περνάμε τώρα στο κλείσιμο λογαριασμών του Άρτεμις. Ποιοι είναι, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, ένας κατά, μία αποχή. Σχέδιο ψηφίσματος. Τώρα άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 19 υπέρ, ένας κατά μία εποχή. «22 λοιπόν για την κοινή δράση Clean Sky» θα υπάρξει και μια προφορική τροπολογία που θα ψηφίσουμε μετά. Τώρα την απαλλαγή ηλεκτρονικά. 19 υπέρ, ένας κατά μία εποχή. Κλείσιμο των λογαριασμών λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 22 υπέρ, 1 κατά, μία αποχή. Καμία αποχή μάλλον εδώ. Τώρα σχέδιο ψηφίσμα ή μάλλον στην προφορική τροπολογία De Jong. Διάρσεως των χειρών ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τελική ψήφος ηλεκτρονικά. Τέλος. 22 υπέρ, ένας κατά, καμία αποχή. 23 τώρα. IMI, κοινή δράση. Έχουμε πάλι προφορική τροπολογία Πρώτα όμως ψηφίζουμε την απαλλαγή ηλεκτρονικά. Τέλος. 19 υπέρ, ένας κατά καμία αποχή. Ε, πρόταση απόφαση για το κλείσιμο των λογαριασμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο 20 υπέρ, ένα κατά καμία αποχή. Προφορική τροπολογία De Jong. Σηκώστε τα χέρια σας. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Και τώρα ηλεκτρονική ψήφος για το τελικό ψήφισμα. Τέλος. 19 υπέρ, ένας κατά καμία αποχή. Τώρα λοιπόν φτάνουμε στο 24. για το ίτερ και την πυρηνική σύνδεξη. Έχουμε και εδώ προφορική τροπολογία του Ντεγιόν. Πρώτα ψηφίζουμε την πρόταση απαλλαγής. Τέλος. 20 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Πρόταση ψηφίσματος για το κλείσιμο τώρα, υπέρ, τέλος. 21 υπέρ 2 κατά καμία αποχή. Τώρα σηκώστε τα χέρια σας για την τροπολογία De Jong, ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονική ψήφος. Τελική. 19 υπέρ, τρεις κατά, καμία αποχή. Και φτάνουμε τώρα στο Ζέζαρ. Η Επιτροπή Μεταφορών έχει καταθέσει τις τροπολογίες 3, 4, 6 και 9 που ήδη περιλαμβάνονται στο κείμενο. Θα θέσουμε πρώτα σε ψηφοφορία την πρόταση απαλλαγής. Ψηφίζουμε. Τέλος. 21 υπέρ, 1 κατά, 1 απέχει. το κλείσιμο των λογαριασμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 23 υπέρ, ένας κατά, καμία αποχή. Τώρα ερχόμαστε στις τροπολογίες. 1, 2, 7, 8 και 5. Ομαδών, εφόσον συμφωνείτε. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ, σηκώστε τα χέρια σας. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Παράγραφος 10. Προφορική τροπολογία de Jong. Υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τελική ψήφος. Τέλος. 22 υπέρ. Ένας κατά. Καμία αποχή. Αυτά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο εισηγητή για την πολλή δουλειά την οποία έκανε. χάρη στην συνεργασία όλων προχωράμε πολύ γρήγορα, σχεδόν μισή ώρα νωρίτερα. Εκπερνάμε λοιπόν με τη γνωστή μας ταχύτητα στο επόμενο σημείο. Για μια στιγμή να μην κάνω λάθος. Ευχαριστώ και τη γραμματεία για την συνδρομή της. Το επόμενο λοιπόν θέμα είναι η έκθεση Ριβελίνη απαλλαγή προς το Συμβούλιο. Θα προχωρήσουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων για την απαλλαγή του προϋπολογισμού του Συμβουλίου. Ψάχνω να βρω τα έγγραφά μου. Έχει υπάρξει και αλληλογραφία επιστολική όπως γνωρίζετε ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και την Επιτροπή μας. Για μια στιγμή διακόπτει ο Πρόεδρος. Inderdaad, we hebben ehm, ehm, Έχουμε λοιπόν ως Επιτροπή λάβει μια επιστολή από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και Το Συμβούλιο μας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, ε, μας έστειλε βέβαια και έγγραφα, κυρίως όσον αφορά την ε, οικονομική κατάσταση από το 2009 τις δηλώσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου, τη συνεργασία για το 2009 με, τους, με τον εσωτερικό έλεγχο. Όμως ο δικός μας ο κατάλογος ερωτημάτων δεν απαντήθηκε και στις 2 ε, Μαρτίου εγκρίθηκε ένα μνημόνιο συναντήληψης που αφορά στις ε, σχέσεις ανάμεσα στο ε, Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και αντικείμενο έχει την απαλλαγή. Αυτό λοιπόν το θέμα θα το εξετάσουμε τώρα. Ο εισηγητής κύριος Ριβελίνη έχει το λόγο και εντωμεταξύ ε, φαντάζομαι ότι θα έχετε συζητήσει με κάποιους αρμόδιους και ε, θεωρώ ότι μπορείτε να μας ενημερώσετε. Γιατί... Συζητάμε σήμερα ένα ντοσιέ πολύ σημαντικό πριν από την ψηφοφορία αύριο και αφορά στην απαλλαγή του Συμβουλίου. Γνωρίζετε, σας έστειλα τον κατάλογο ψηφοφορίας, είναι να καθυστερήσουμε την απαλλαγή του Συμβουλίου και έχω τρεις βασικούς λόγους που ενέκρινε η ομάδα μου. Πρώτος λόγος, το Συμβούλιο δεν δέχτηκε καμία από τις προσκλήσεις μας να συναντήσει την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου ή τον εισηγητή, δηλαδή εμένα, για να συζητήσουμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το 2009. Δεύτερος λόγος, το Συμβούλιο αρνήθηκε να δώσει γραπτή απάντηση στο ερωτηματολόγιο το οποίο έστειλε ο εισηγητής στις 14 Δεκεμβρίου του 2010. Τρίτος λόγος, το Κοινοβούλιο δεν έλαβε τα βασικά έγγραφα του Συμβουλίου όπως ας πούμε τον πλήρη έλεγχο των ε, εκτελέσεων του προϋπολογισμού. Εγώ δεν θέλω να σταθώ ε, στην επιλογή μου ε, αλλά και άλλων ομάδων να μην χορηγήσω την απαλλαγή. Η πολιτική κρίση του κάθε βουλευτή θα εκφραστεί αύριο με την ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή ή όχι. Πιστεύω ότι η τοποθέτησή μου μπορεί να είναι χρήσιμη κυρίως ε, για τη συζήτηση, εάν δηλαδή την τοποθετήσουμε σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Για να το πω απλά δηλαδή στο τι συνέχεια θα δώσουμε στην ψηφοφορία αύριο. Πρέπει λοιπόν εμείς να αναρωτηθούμε σε αυτήν τη διαδικασία απαλλαγή ποιος είναι ο ρόλος μας ως Επιτροπή Προϋπολογισμών και πιο συγκεκριμένα τι διέξοδο έχουμε από, την, από αυτό το θεσμικό τέλμα στο οποίο έχουμε πέσει εδώ και μερικά χρόνια. Να είμαι τώρα σαφέστερος και να υποδείξω ποιες είναι οι πιθανές λύσεις Πρώτη λύση και μετά θα ακολουθήσουν σχόλια. Πρόκειται για τη λύση που έχει τη νομική βάση στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την απαλλαγή του 2008 και που προβλέπει την αποστολή των εξής εγγράφων. Λογαριασμοί του προηγούμενου οικονομικού έτους ε, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 2. Προϋπολογισμός με ενεργητικό και παθητικό. Τρίτο, ετήσια έκθεση για τη διαχείριση του προϋπολογισμού και δημοσιονομική διαχείριση. Τέσσερο, ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή. Και θα πρέπει να περιλαμβάνει και μία προφορική παρουσίαση κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής κατά τη διαδικασία της απαλλαγής. Δεύτερη λύση. Το Συμβούλιο υπόκειται σε μια διαδικασία σαν αυτή όλων των υπολείπων θεσμικών οργάνων. Οπότε το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται συστάσεις από το Συμβούλιο. Τρίτη λύση έχει να κάνει με τη διαθεσμική συμφωνία που προβλέπει διάφορες φάσεις και διαδικασίες που πρέπει να γίνουν σεβαστές. και που μειώνουν βέβαια τις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής υπέρ της διάσκεψης των Προέδρων και της Επιτροπής Θεσμικών Υποθέσεων. Όπως είπατε υπάρχουν καινούρια. Ο κύριος Δεμπισιέ, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου, στις 16 Μαρτίου, ανακοινώνει αυτός ο κύριος ε, στον, στον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βέλε, να προχωρήσει με την τρίτη λύση, δηλαδή με τη διαθεσμική συμφωνία. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την τελευταία επιστολή, προσωπικά θεωρώ ότι καμιά από τις τρεις προτάσεις μας ικανοποιεί απόλυτα, διότι φυσικά δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Χρειάζεται όμως να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για να σώσουμε το καλό όνομα των θεσμικών οργάνων. Ένα λοιπόν πρώτο αποτέλεσμα κοινοβουλευτικά το έχουμε βρει στο βαθμό που η Επιτροπή μας έχει ξαναβρει τον κεντρικό της ρόλο. Πρέπει θεωρώ να βασιστούμε στο ψήφισμα του περασμένου Ιουνίου και ζητώ από εσά συνάδελφοι να εκφραστείτε σχετικά και να ξεκινήσουμε μία συζήτηση ώστε να έχουμε στο μέλλον μία κοινή θέση. Εγώ στο τέλος θα προτείνω μία λύση αφού σας ακούσω. Και αυτό για να μην εκφραστώ εδώ με μία γραμμή αδιάλακτη ή προδικασμένη. Αλλά δεν πρέπει όμως να προδικάσουμε και στο Συμβούλιο ένα ειδικό καθεστώς. Σας ευχαριστούμε κύριε Ριβελίνη. Μέχρι τώρα δεν ήταν να ζητάει κάποιος το λόγο. Α, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η κυρία Γιάλα Σέντερ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ριβελίνη για όλη του την προσπάθεια συμπιαλλαγής και με την Ουγγρική Προεδρία και με τους σκεώδεις εισηγητές. Εγώ θα έλεγα ότι εμείς φέτος στην αντίστοιχη φάση της διαδικασίας έχουμε κάνει ένα πίσω γύρισμα. Είμαστε ένα βήμα πίσω από ό,τι ήμασταν πέρυσι με την Ισπανική Προεδρία. Πέρυσι έστω και αν ακολουθήσαμε διαδικασίες που δεν ήταν παγιωμένες, είχαμε κάποιες απαντήσεις τουλάχιστον φέτος, δεν είχαμε καν αυτή τη συνεργασία. Ελπίζω αυτή η Κομισιόν, αυτή συγγνώμη η Επιτροπή να πετύχει την αναβολή της απαλλαγής του Συμβουλίου. Βρισκόμαστε σε μια κριτική φάση. όπου θα πρέπει να εκπληρώσουμε αυτό το οποίο ορίζει συνθήκη. Δηλαδή ότι το Κοινοβούλιο αποφασίζει για τα άλλα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς. Μας αναγνωρίζετε. ο αποφασιστικός μας ρόλος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει οριστικά. Θα πρέπει να πετύχουμε την αναβολή και επικυρώνω όλα όσα μας είπε ο κύριος Ριβελίνη. Υπάρχει Δεν έχει μάλλον δοθεί απάντηση σε όλα όσα έχει ρωτήσει το Κοινοβούλιο μέχρι σήμερα. Πρέπει να τελειώνουμε, να δοθούν απαντήσεις. Και μέχρι την Ολομέλεια να ξεκαθαρίσουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και να δούμε τι θα κάνουμε με το Συμβούλιο, διότι το Συμβούλιο κατά την άσκηση του έργου του εργάζεται, έχει διοικητικές δαπάνες και υπάρχουν λειτουργικές δαπάνες πολύ σημαντικές και επειδή αποτελούν τμήμα του κοινοτικού προϋπολογισμού θα πρέπει να εγκρίνονται ως προς τη διαχείρισή τους και αυτό ήθιστε με όλα τα θεσμικά όργανα. Πρέπει να πετύχουμε να ολοκληρώσουμε την απαλλαγή όπως κάναμε και με όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Και να μην καταλήξουμε σε μια ανώμαλη κατάσταση λόγω αυτής της πολεμικής. Προτιμώ να αναβάλουμε την ψηφοφορία, όπως είπε και ο κύριος Ριβελίνη, και να πετύχουμε μια πλειοψηφική υποστήριξη. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκάια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι τώρα καθόλου σίγουρος ε, σχετικά με όλο αυτό το ιστορικό που οδήγησε στην ανταλλαγή επιστολών. Διότι κατά τη δική μου άποψη τη θέση της Επιτροπής την είχαμε διευκρινίσει, επαρκώς τουλάχιστον. Και μάλιστα... Ε, η θέση ήταν τόσο σαφής που πλέον δεν γνωρίζω ε, πάνω σε ποια βάση αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Συμβουλίου να θέσει το θέμα της διοργανικής συμφωνίας. Εγώ ε, μέχρι τώρα είχα καταλάβει ότι η θέση της Επιτροπής είναι ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να χορηγήσει την απαλλαγή ε, σε εκείνα τα θέματα που αφορούν στον κοινωνικό προπολογισμό, ότι δεν αμφισβητεί αυτή τη διαδικασία. Και αν ισχύει αυτό, τότε τι να διαπραγματευτούμε. Μια διοργανική συμφωνία, η οποία είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων από τη διάσκεψη των προϊόντων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα τελείω διαφορετικό αποτέλεσμα. Εγώ λοιπόν δεν κατάλαβα ποιο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα, ποιος ε, εγκρίνει αυτό το αποτέλεσμα σε αυτή την Επιτροπή και τι τελικά θα αποκομίσουμε. Η στάση αυτής της Επιτροπής θα έλεγα ότι είναι σαφής, ότι εμείς ε, ερμηνεύουμε τη συνθήκη ε, με τον έννοια ότι ε, η Επιτροπή Προλογισμών είναι η αρμόδια επιτροπή που χορηγεί την απαλλαγή. Το Συμβούλιο επιμένει στην αμοιβαιότητα, πράγμα που μέχρι τώρα είχαμε απορρίψει και αν τελικά υπάρξει μια διοργανική συμφωνία, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή πέρα από αυτά που ήδη αναφέρονται στη συνθήκη. Πρόεδρος, ε, πολύ ενδιαφέρουσε παρατήρηση. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ε, κύριε Πρόεδρε, εγώ από πλευρά περιεχομένου ε, συμφωνώ με τον κύριο Γκάγια και γι' αυτό το λόγο και εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό να έχουμε ε, αναβολή και όχι χορήγηση απαλλαγή Πράγματι, τα ερωτήματα που θέσαμε δεν απαντήθηκαν επαρκώς. Η συμφωνία συναντήληψη με την Κορεπέρ δεν μα ικανοποιεί και έχω την εντύπωση ότι επανερχόμεθα στη συζήτηση τη τελευταίες εβδομάδες όπου είχαμε συγχυτή τον κύριο Ζόνενγκάρτ και κατόπιν τούτου εγώ νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε αναβολή. Όσον αφορά τα αιτήματα του Συμβουλίου προς εμάς πρέπει να τα ελέγξουμε ένα προς ένα. Δεν μπορούμε να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως και να κλείσουμε την πόρτα. Όμως η προϋπόθεση για διαπραγμάτευση είναι η σαφή διευκρίνηση του ερωτήματο ποιο είναι ο αρμόδιο. Όπως είπε και ο κύριο Γκάιερ, η συνθήκη είναι σαφή στο θέμα αυτό. Αν λοιπόν το Συμβούλιο αμφισβητεί αυτό το θέμα, παρακαλώ και τον εισηγητή μα, το άρθρο 256 του κανονισμού μα, ε, να το εκμεταλλευτούμε και να καταφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πράγματι ε, θα πρέπει να καταφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην περίπτωση κατά την οποία ε, το Συμβούλιο αμφισβητεί την αρμοδιότητά μας ως Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Αυτό το αναφέρει όπως σας είπα συνθήκη. Πρέπει λοιπόν να το ελέγξουμε αυτό και να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά διότι φοβάμαι ότι το Συμβούλιο δεν κάνει κανένα βήμα προς τα μπρος αλλά το αντίον κάνει βήματα προς τα πίσω. Κύριε Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι όσον αφορά το τι θα κάνουμε με το Συμβούλιο, η αναβολή της αποβολής, της απαλλαγής, αυτό είναι σωστό, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε στο μέλλον. Πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει λιγάκι ως προς την ανταλλαγή επιστολών ε, την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη. Και πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ ε, δεν το κατάλαβα κιόλας. Δηλαδή, ε, και εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτό οφείλεται στο ότι ε, δεν ξέρω πάρα πολύ καλά αγγλικά και το μετάνιωσα που στο μάθημα των αγγλικών στο σχολείο δεν πρόσεχα αρκετά. Αλλά για όλου του λόγου, εμάς πάση περιπτώσει, πήρα τηλέφωνο τον κύριο Βέλε την Παρασκευή και ο κύριο Βέλε μου είπε ότι είτε θα δεχτείτε αυτό το οποίο ε, προτείνει η Επιτροπή Προϋπολογισμών είτε θα κάνουμε κάτι διαφορετικό ε, και θα είναι πιο χρονοβόρα αυτή η διαδικασία και θα διαπραγματευτούμε την αμοιβαιότητα. Αυτή λοιπόν ε, ήταν η πρόταση και το Συμβουλίο επέλεξε τη διοργανική συμφωνία. Και ομολογώ ότι αυτό με εντυπωσίασε. Ε, κοιτάξτε, ε, σε αυτό το θέμα νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν λέω ε, το σημείο 8 να το εμπλουτίσουμε με μια προφορική τροπολογία και να πούμε θεωρεί ε, η διοργανική συμφωνία για την απαλλαγή του Συμβουλίου δεν είναι απαραίτητη. Κάτι τέτοιο περίπου στη διατύπωση να λάβουμε θέση. Γιατί και εγώ νομίζω ότι τη διοργανική συμφωνία δεν την χρειαζόμαστε. Και εάν την πάρουμε τελικά εκεί μπορεί να αναφέρονται πράγματα που δεν μας αρέσουν. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι το Συμβούλιο βεβαίως ε, βρίσκεται εμπλεγμένο σε σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή ε, το Συμβούλιο ασχολείται με τον κοινωνικό προπολογισμό και τα κράτη με μελη ασχολούνται με τους γεωργικούς προϋπολογισμούς. Εγώ λοιπόν δεν έχω καμία όρεξη να δεχθώ εκβιασμούς. Θα ήθελα λοιπόν αύριο να ξεκαθαριστεί το θέμα και γι' αυτό εγώ προσπάθησα να σας προειδοποιήσω και είπα προφορική τροπολογία στο σημείο 8, άσχετα που θα μπει τώρα, δεν έχει καμία σημασία, απλά να ε, καθιστούμε σαφές ότι η διοργανική συμφωνία δεν απαιτεί ε, να υπάρχει ξεχωριστή συμφωνία. Και είμαι ευγνώμων στο Γενικό Γραμματέα τον κύριο Βέλε, διότι θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες για ε, να λυθεί το θέμα. Θα δούμε βέβαια πώς θα προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι το Συμβούλιο δεν προσπάθησε καθόλου, δεν έκανε τίποτα. Και τώρα να θέλει να κάνει κάτι το Συμβούλιο όσον αφορά ε, στο Κοινοβούλιο, αυτό είναι άδικο και εμείς έτσι και αλλιώς ε, θέλουμε απλά το ε, Συμβούλιο να δέχεται αυτά που προτείνουμε και τα ορίζουμε. Δεν θέλουμε τίποτα πέρα από αυτό. Πάντως για μας σας λέω το θέμα θα είναι αρνητικό, θα πάρουμε λιγότερα ε, και θα ήταν και ένα λάθος μήνυμα που θα εκπέμπαμε προς την κοινή γνώμη, προς τα έξω. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Είπατε ότι ε, λυπάστε πάρα πολύ που δεν ήσταν καλή μαθήτρια στο σχολείο. Μα πώς γίνεται το εδώ, είστε καταπληκτικοί προσέχτες συνέχεια και στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο. Δεν αμφισβητεί κανείς την επιμελιά σας. Πάντως ε, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια ειδική τροπολογία για τη διοργανική συμφωνία. Πρόκειται για ένα νέο στοιχείο στη συζήτηση. Θέλει κάποιος να λάβει το λόγο. Αν όχι θα το δώσω στον εισηγητή. Ε, η κυρία Αγιά Λάσεν, ε, παρακαλώ. Αυτό το οποίο λέει η κυρία Γκρέσλερ είναι απόλυτα καινούριο. Αυτό το οποίο μας δέσμευσε τον κύριο Ριβελίνη και εμένα. Τι λέμε, ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια εστίαση που έχουμε με τα άλλα θεσμικά όργανα και αυτό ήταν σαφές. Εγώ τώρα δεν ξέρω Δεν ξέρω γιατί αν είμαστε κατά Δηλαδή ο κύριος ε, Κλάους Βέλε αποφάσισε άλλα πράγματα και εμείς υποβάλλουμε εδώ μια προφορική τροπολογία εντελώς αντίθετη. Θα ήταν καλύτερα λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Κλάους Βέλε πρώτα. Και δεν καταλαβαίνω εγώ, ενώ εργάστηκε καλά, να θα πρέπει εμείς να, του, να ανοίξουμε τα χαρτιά μας ε, στο Συμβούλιο δείχνοντάς του κατευθείαν ποια είναι η στρατηγική μας. Εγώ θα προτιμούσα την παρανομή της ψηφοφορίας να αποφασίσουμε σήμερα αλλά ε, δεν ξέρω γιατί θα ήταν καλύτερα να ακούσουμε το γενικό μας γραμματέα αν έχει αποφασίσει ή αν έχει αποφασίσει κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ πάντως, όπως λέει και ο κύριος Ριβελίνη, ότι αντιμετωπίζουμε το Συμβούλιο όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα. Εγώ δεν θα ήθελα να κλείσουμε μία πόρτα γιατί δεν ξέρω πραγματικά που θα μας πάει. Πρόεδρος, κοιτάξτε, έχουμε χρόνο. Η ψηφοφορία θα είναι αύριο και η κυρία Κρέσλε θα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει προφορική τροπολογία. Νομίζω ότι αυτό είναι δικαίωμά τη ε, ως ε, βουλευτής έχει αυτή τη δυνατότητα ε, μπορεί κανείς να ξαναδεί το θέμα με την άλλη κυρία Κρέσλε. θέλετε να λάβετε το λόγο κοιτάξτε αν θέλουμε την πεπατημένη Υπάρχουν δύο δυνατότητε. είτε η πεπατημένη είτε η διοργανική συμφωνία. Νομίζω αυτό αναφέρεται ρητά στην επιστολή. Ε, και εγώ είμαι υπέρ τη πεπατημένη. Εμεί ε, τι επιτιμούμε να έχουμε. Εγώ θέλω την πεπατημένη, τη συνήθεια δηλαδή δικασία και καμία διοργανική νέα συμφωνία. Γιατί με την συνήθεια δικασία δεν χρειαζόμαστε διοργανική και αυτό θέλω να φανεί με απόλυτη σαφήνεια. Εγώ επιθυμώ να υπάρχει μια απόλυτα κανονική ε, διαδικασία με το Συμβούλιο. Ε, δεν θέλω να υπάρχουν ε, μισέ λύσει, να παρατηθούμε από κάτι, το Συμβούλιο να κάνει κάτι άλλο, να μην κάνει καθόλου κάτι άλλο, να προβεί ίσω σε συμφωνία των κυρίων για την απαλλαγή, όπου θα αναφέρεται κανεί για θα βλάψει τον άλλον. Αυτή κατ' ουσίαν είναι η κρυφή επιτιμία του Συμβουλίου. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με όλα αυτά. Γι' αυτό σα λέω ότι εγώ είμαι περισσότερο υπέρ του να ε, προσθεθεί αυτή η πρόταση όπου θα καθιστούμε απόλυτα σαφές το τι επιθυμούμε. Γιατί, ε, να το πω έτσι κάπως πιο προσεκτικά, ε, δεν έχουμε όλους τους ίδιους στόχους εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε. Και εγώ δεν χρειάζεται αν θέλετε να κάνω τίποτα και εγώ μπορώ να κάτσω και να παρατηρώ απλά τι γίνεται. Ο κύριος Ριβελίνη. Εγώ έχω την τάση να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Και φυσικά η συζήτηση που γίνεται εδώ και μήνες, γιατί μήνες κράτησε αυτή η συζήτηση, έχει θέσει το Κοινοβούλιο σε μια κεντρική θέση. Επίσης, έδειξε προς το Συμβούλιο ότι υπάρχει μία συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων ώστε να καταστεί σεβαστός αυτός ο κεντρικός ρόλος του Κοινοβουλίου και εμείς με αυτήν την τελευταία επιστολή που λάβαμε ε, καταλήγουμε σε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι ικανοποιητικά σήμερα για τους βουλευτές οι ψηφοφορίες και οι συμφωνίες που συνάψαμε με άλλους συναδέλφους για αύριο για την ψηφοφορία ε, είναι καρπός, μάλλον καλύτερα αντικατοπτρίζει τις θέσεις όλων των βουλευτών. Εγώ σας παρουσίασα τις τρεις λύσεις, δεν υπάρχουν άλλες. Τρεις λύσεις για να βγούμε από την κρίση η τροπολογία αύριο εκ μέρους της κυρίας Γκρέσελ θα αποτελεί την επικύρωση της θέσης μας. Έχουμε καιρό ως αύριο για να το συζητήσουμε και για να το σκεφτούμε. Η αλήθεια όμως ποια είναι και πρέπει να τη λέμε γιατί αλλιώ θα ξεχάσουμε όλα τα βήματα τα οποία κάναμε μέχρι τώρα. Είναι λοιπόν η θέση μας. το Κοινοβούλιο να γίνεται σεβαστό από τα άλλα όργανα. Και αυτή η πεποίθηση των βουλευτών για τον ρόλο του Κοινοβουλίου μας καθιστά σεβαστούς έναντι του Συμβουλίου. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο, πάντοτε με την ίδια αυστηρότητα, χωρίς βέβαια ποτέ να σταματήσουμε να ακούμε η κουλτούρα του διαλόγου πρέπει να είναι σημαντική σε μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αύριο η ψηφοφορία είναι αρκετά σαφής. Θα συζητήσουμε εμεί σήμερα για αυτή την τροπολογία που απλώς θα επικυρώσει αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Το λέω προς τη συνάδελφα Αγιάλα. Πολύ ωραία λοιπόν, λέει ο πρόεδρος, ε, μήπως υπάρχει κάποιος άλλος, επιθυμεί κάποιος άλλος ε, να λάβει το λόγο. Νομίζω ότι στην αίθουσα είχα, έχουμε και εκπροσώπους του Συμβουλίου, οι οποίοι φαντάζομαι παρακολούθησαν, ε, τα όσα ελέγχθησαν, τα κατάλαβαν και νομίζω ότι κατέστη απόλυτα σαφής ε, ε, η ενιαία στάση, η ομόφωνη στάση ε, που υπάρχει στο Συμβούλιο. Αύριο λοιπόν θα ψηφίσουμε για την απαλλαγή. Κατόπιν τούτου πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, που είναι το επαριθμόν 27 και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Πρόκειται για το έγγραφο 815 ε, του 2010 της Κομισιόν ε, πρόκειται για τους ε, κανόνες ε, σχετικά με τον ετήσιο προπολογισμό, ένα έγγραφο της 22ης Δεκεμβρίου. Διαδικαστικό, παρακαλώ. Θα ψηφίσουμε αύριο θα, ψηφίσουμε αύριο. Αλλά εγώ θέλω όμως να συζητήσουμε αύριο και με τον κύριο Ριβελίνη για το θέμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Δεν το έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη, αλλά ούτε και αύριο. Και επειδή αύριο θα το ψηφίσουμε, εγώ θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Ριβελίνη για αυτό το θέμα, αν φυσικά είναι δυνατόν. Ναι, εντάξει, να το κάνουμε αύριο. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε αύριο, λίγο πριν από την ψηφοφορία, να συζητήσουμε για την άποψη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Κοιτάξτε, τώρα είμαστε μισή ώρα μπροστά. Έχουμε δηλαδή, αν θέλετε, έχουμε μια μισή ώρα για την έκθεση Ριβελίνη Γκρέσλε και δεν τα χρειαστούμε κατά πάσα πιθανότητα αυτά τα 90 λεπτά. Ε, μέχρι τις 5.30 ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε και ένα διάλειμμα και μπορείτε εσείς να μιλήσετε τότε αν θέλετε για την ΟΚΕ. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 27. Είχα ήδη αρχίσει, είχα ξεκινήσει ε, να κάνω μία μικρή εισαγωγή. Ας το κλείσουμε αυτό το θέμα και μετά θα λάβετε εσείς το λόγο για την ΟΚΕ ανάλογα με το πόσο χρόνο θα έχουμε στη διάθεσή μας για να μιλήσουμε με τον κύριο Εγκβίρντα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια πολύ σημαντική πρόταση αυτή τη ε, Κομισιόν, την οποία ε, καλούμεθα να συζητήσουμε. Είναι ένα νέο έγγραφο ε, τη Κομισιόν, το οποίο αντικαθιστά δύο παλαιότερα. Ο κύριο Ριβελίνη και η κυρία Γκρέσλε συνέστησαν ομάδα εργασία που συναντήθηκε επανειλημμένα για να προετοιμάσει αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που σας είπα. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα πρόκειται για μια συζήτηση ε, που προβλέπεται στις 13 και 14 Απριλίου σχετικά με τον προπολογισμό. Ε, σε αυτή τη συζήτηση είναι, είμαστε προσκεκλημένοι και εμείς. Ε, θα ήθελα όμως καταρχήν να δώσω το λόγο Βελίνη, ο οποίος θα λάβει το λόγο εξ ονόματός μας. Ε, της Επιτροπής μας. Μπορείτε λοιπόν κύριε Ριβελίνη αν θέλετε να μας παρουσιάσετε το έγγραφο. Βεβαίως και θα λάβει το λόγο κατόπιν η κυρία Γκρέσλε και ίσως και όποιος άλλος επιθυμεί. Ο κύριος ε, Ριβελίνη. Συζητάμε εδώ το έγγραφο που παρουσιάστηκε για την μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού. Εγώ δεν θέλω να κλέψω χρόνο τη συζήτηση. Και θα ήθελα όμως να δώσω και τον επαρκή χώρο στην κυρία Γκρέσλερ για να μπορέσει να μας εκφράσει αναλυτικότερα τις πιο σημαντικότερες αλλαγές. Θα περιοριστώ μόνο σε μία εισαγωγή και θα κοιτάξω το συντομότερο δυνατό να αναφέρω τη χρήση των δημοσιονομικών μέσων. Παραπέμπω στο έγγραφο εργασίας για περισσότερες λεπτομέρειες. Στη γενική πλαισίωση όπως γνωρίζετε στο 0815 μετά από έντονες συζητήσεις ε, τον Δεκέμβρη του 2010 συμπεριλαμβάνει και τη διαδικασία της Λισαβονα ε, και την περασμένη διαδικασία και τροποποιεί πάνω από τα μισά από τα 200 άρθρα. Άμεση επίπτωση αυτής της επιλογής που είναι πολύ ορθή και που τη θέλαμε είναι η άσκηση εκ μέρους του Κοινοβουλίου της συναπόφασης. Δικαίωμα που για τον δημοσιονομικό κανονισμό ήδη ισχύει από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Διαφορετικές όμως ήταν οι άτυπες συζητήσει που είχαμε στην ομάδα εργασίας όπου τονίστηκαν ε, αντιλήψεις ε, και άλλαγες που θέλουν να εισάγουν στο δημοσιονομικό κανονισμό. Και εμείς από τη μεριά μας όμως σταθήκαμε στα εξής. Οι ουσιαστικές αλλαγές για τις επιστροφές στον προϋπολογισμό και η περιφρούρηση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου ως, κλαδ, ως αρχή του προϋπολογισμού. Δεύτερο, η νέα αντίληψη του ρίσκου και του ανεκτού λάθος. 3. Εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού και πιο συγκεκριμένα η επανοδιοργάνωση των τωρινών ε, μεθόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και άμεση και έμεση διαχείριση. Επίσης, ανάθεση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στην ΕΤΕ. Τέσσερα, το θέμα των δημοσιονομικών μέσων έτσι όπως περιγράφονται από την πρόταση της Κομισιόν, μελλοντικός ρόλος της ΕΤΕ και των άλλων δημοσιονομικών οργάνων. Έξι, οι, ανα, οι ανατιθέμενες πράξεις για την ανάθεση εξουσιών στην Κομισιόν για την πρόταση αναθεώρησης των εκτελεστικών λεπτομεριών του κανονισμού. Γενικές ε, τώρα, ε, γενικές θεωρήσεις για αυτά που σας είπα. Όπως σας είπα πριν, είναι ποικίλε και σύνθετες οι διάφορες θεματικές και πάντοτε έχουν να κάνουν στο με τον προπολογισμό αφενός και απετέρου ε, συνδέονται με τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Εμείς ήδη θυμήσαμε στις προηγούμενες συνεδριάσεις το θέμα του ανεκτού λάθους. Θεματική που τη γνωρίζουν ήδη οι συνάδελφοι οι οποίοι παρακολουθούν αυτήν είναι μέλη της Επιτροπής πολύ πριν από μένα. Και η πρόταση της Επιτροπής αντιμετωπίστηκε ε, σχετικά επιφανειακά και που μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο έγγραφο εργασίας. Προτείνουμε λοιπόν εμείς να τροποποιήσουμε την πρόταση της Κομισιόν, ούτως ώστε ο αποδεκτός κίνδυνος σφάλματος να γίνει ένα μέσο διαχείρισης που θα εκτιμά τους διαχειριστές πολιτικούς ε, ε, τρόπους. Και έτσι η Κομισιόν θα μπορεί να παρακολουθεί από κοντά τον έλεγχο των προγραμμάτων και να αντιδρά αναλαμβάνοντας διαφορετικά μέσα περισσότερους ελέγχους, ε, ενίσχυση των προγραμμάτων κλπ. Χρειάζεται να γίνεται επαλήθευση ένα ταμείο και ένα κράτος μέλος αλλά για τη σωστή διαχείριση των κονδυλίων και σε τέτοιες δύσκολες στιγμές σαν αυτές θα έπρεπε να τη χάνουν της απαραίτητης σημασίας. και μέλη του γραφείου του αρμοδίου επιτρόπου και η Κομισιόν η ίδια εξέφρασαν τις ανησυχίες τους και πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Ε, για τη χρήση πάντως των δημοσιονομικών μέσων πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό. Και να επανέλθω τώρα στην αρχική ε, τοποθέτηση. Για τα χρηματοπιστωτικά μέσα πριν αρχίσω να κρίνω να σας πλαισιώσω λίγο την κατάσταση. Η πρόταση της Κομισιόν αφορά σε δύο άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού, το 130 και το 131 και τρία άρθρα των εφαρμοστικών λεπτομεριών. Από το, από το συγγνώμη, 39 γάμα στο 39 ε. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό ε, και ευρύ. Πρόκειται για μέτρα χρηματοπιστωτικής υποστήριξης της Ένωσης που βαρύνουν τον προϋπολογισμό και στοχεύουν σε ένα ειδικό ε, σημείο με μετοχικούς δανισμούς ή άλλα μέσα ρίσκου που συνδέονται με επιδότηση. Τα δημοσιονομικά μέσα σε πολλές περιπτώσεις είναι πολιετή προγράμματα και για να συλλέξει ταμεία η Κομισιόν έχει την πρόθεση να εκδώσει τα project bond η πρόταση λέει ότι αυτός ο οποίος θα ασχολείται με την εφαρμογή θα είναι η ΕΤΕ η οποία θα αντιμετωπίζεται με ειδική μεταχείριση ως όργανο βάση της συνθήκης και θα εξαιρείται από τις διαδικασίες διαγωνισμού ανάθεσης δημοσίων έργων και από τις ε, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για διαδικασίες χορήγηση επιδοτήσεων. Χρειάζονται τώρα περαιτέρω διευκρινήσεις από την Επιτροπή όσον αφορά στην σελεκτικές διαδικασίες. Το να μπορεί κανείς τώρα να δίνει σε υπεργολαβία την εκτέλεση σε μία θηγατική και κάτω από τη δική της ευθύνη δεν θα βρίσκεται πλέον αυτό στα χέρια του Κοινοβουλίου διότι θα είναι εντελώς ανεξάρτητο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι για να μην συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζονται έλεγχοι διότι οι μηχανισμοί ελέγχου δεν θα βρισκόταν πλέον στα χέρια του Κοινοβουλίου αλλά θα οριζόντουσαν στην απόφαση ανάθεσης και στο πλαίσιο των συμφωνιών που θα έχουμε διαπραγματευτεί με την ΕΤΕ, άρθρο 39 39Γ, στην παράγραφο 1 και 2. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε σημαντικά τις διατάξεις που προτείνονται και αυτό προτείνοντας να εναρμονίσουμε ε, τους κανόνες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη και να αποφύγουμε τις αντιφάσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και μία προσέγγιση ε, των πολιτικών προτεραιοτήτων. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα ειδικό καθεστώς ε, και αυτό βάσει των ε, όσων ορίζει η συνθήκη. Θα πρέπει να εγγυθούμε οι μελλοντικές αναθέσεις να γίνονται με μια ειδική νομική βάση και να διατηρείται η αρμοδιότητα της Επιτροπής ως προς την εκτέλεση. Οι τελικές ε, θεωρήσεις μου είναι η εξής. Η πρόσταση της Κομισιόν να χρησιμοποιήσει μέσα που θα τις διαθέτει η χρηματοπιστωτική αγορά, αυτό θα πρέπει να το δούμε με καλό μάτι. Πόσο μάλλον στο τωρινό πλαίσιο των, της οικονομικής κατάστασης. Σε μία φάση που τα κράτη υποφέρουν ε, λόγω του κυρίαρχου κρέους και όπου αμφισβητείται η χρηματοδότηση των κοινοτικών πολιτικών και συζητάμε όλη την αναθεώρηση των ιδίων πόρων, ο πολλαπλασιωστικός παράγοντας που μας παρέχεται από τη χρήση των δημοσιονομικών μέσων θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να ενισχύσει την αδύναμη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ταυτόχρονα θα εντατικοποιούσε και τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση χρηματοδότησης. Επίσης, άλλα που θα πρέπει να στα θα πρέπει να εμπαθύνουμε επιπτώσεις ε, στις ε, προοπτικές ε, του προϋπολογισμού και αλλαγή της οικονομικής governance. Θα ήθελα όμως τώρα να αφήσω το λόγο στην κυρία Γκρέστελ η οποία θα μπορέσει να μας διευκρινίσει καλύτερα άλλα στοιχεία που αφορούν στην άμεση και έμεση διαχείριση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσελ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ριβελίνη και όλους τους ε, συναδέλφους που παρέμειναν εδώ γιατί ε, στην Επιτροπή Προπολογισμού χρειάστηκαν τρία λεπτά για να διάσει αίθουσα. Ε, εδώ όμως βλέπουμε το ίδιο και το εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό. Βεβαίως πάντα ίδιοι είναι αυτοί που παραμένουν. Κοιτάξτε, πράγματι λοιπόν συστήσαμε μία ομάδα εργασία και δεν θέλω να το πείτε παραπέρα, αλλά εμείς ε, πραγματικά ζηλεύουμε το ε, Συμβουλίο γιατί εκεί είναι 26 άνθρωποι και ε, επικρατεί κάπως πειθαρχία αυτού λεχθέντος. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σε δύσκολη κατάσταση γιατί τα κείμενα τροποποιούνται συνεχώς και οποτεδήποτε συμφωνούμε, κάθε φορά που συμφωνούμε σε μια συγκεκριμένη εκδοχή μπορούμε να είμαστε και σίγουροι ότι θα μας υποβληθεί ένα νέο κείμενο. Αυτά τα νέα κείμενα ε, λοιπόν αφορούν ε, το non-paper που προέκυψε μετά το σεμινάριο της ε, Κομισιόν. Το γεγονός ότι έγινε αυτό το σεμινάριο το βρίσκω πολύ σημαντικό. Υπάρχει λοιπόν ένα non-paper για τα χρηματοδοτικά μέσα και για το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Όσον αφορά τώρα την κοινή διαχείριση, τα χρηματοδοτικά μέσα και τη νομική πράξη όπως και τα ΣΔΙΤ, για αυτά θα σας μιλήσω τώρα τα χρηματοδοτικά μέσα και τα ΣΔΙΤ ο συνάδελφο κύριο Ριβελίνη δεν είμαστε αντίθετοι. Το θέμα που τίθεται μόνο είναι πώ θα γίνουν όλα αυτά. Γιατί και στα δύο μοντέλα, όπω και στι ε, κατεξουσιοδότηση πράξη, σε τελική ανάλυση όλα αυτά σημαίνουν ότι το Κοινοβούλιο χάνει κάθε επιρροή στο τι διαδραματίζεται. Τα υπάρχοντα ΣΔΙΤ αυτή τη στιγμή είναι όλες, όλοι οι κανονισμοί του Συμβουλίου. Είναι κανονισμοί του ε, Συμβουλίου. Πρέπει λοιπόν να διορτηθούμε το εξή. Αν επιθυμούμε κάτι τέτοιο, τότε πώ επιθυμούμε να γίνει. Το θέμα δεν είναι αν είσαι υπέρ ή κατά, το θέμα είναι πώς. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με την κοινή διαχείριση. Εκεί επικρατεί και η μεγαλύτερη σύγχυση. Ε, και θα κάνουμε δύο πράγματα. Αφενός θα επεξεργαστούμε την ήδη επεξεργασμένη πρόταση Κομισιόν, πρόκειται για ένα non-paper, όπου θα διερωτηθούμε τι ρόλο παίζει η Κομισιόν στη διαπίστευση. Και οποτεδήποτε υπάρχει διαπίστευση από την Κομισιόν, το θέμα αυτό γίνεται πολύ δύσκολο, γιατί νομίζω ότι η Κομισιόν ε, μας είπε ότι δεν είναι καν σε θέση να το κάνει αυτό και αν έπρεπε να το κάνει το τίμημα θα ήταν ε, αργοπορημένη εκείνη των προγραμμάτων. Και για να μην γίνουν όλα αυτά συμφωνήσαμε να ζητάμε ανάλυση κινδύνου ή να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ε, να προτείνουν στην Κομισιόν να ελέγχει τα συστήματά τους. Άρα δηλαδή και ανάλυση κινδύνων και εκεί ε, έχουμε ειδικού εμπειρογνώμονες. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι είναι μάλιστα προς όφελος της ε, Κομισιόν να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε λοιπόν να προβλέψουμε αυτή τη δυνατότητα ή και να δώσουμε δυνατότητα ε, στο κράτος μέλου να εκτιθεί κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα, δουλεύουμε με βάση το πρώην άρθρο 153β, όπου ε, ίσως τα κράτη-μέλη, αν τελικά αποφασίσουν να παραμείνουν τα πάντα έχουν, εμείς ε, δεν νομίζουμε ότι μπορούν να παραμείνουν ως έχουν, γιατί θεωρούμε ότι τα υπάρχοντα συστήματα πρέπει να βελτιωθούν. Και το ερώτημα ε, μα πού μπορούν να βελτιωθούν. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, τα ερωτήματα που έβαλα στην Κομισιόν ε, δεν απαντήθηκαν από τους 240 μάλιστα εκπροσώπους ε, ελεγκτές κρατών μελών. Και κρίμα, πολύ κρίμα. Ε, θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε μία βελτίωση. Η μεγαλύτερη ασάφεια, κατά την άποψή μου, εξακολουθεί να υπάρχει στα χρηματοδοτικά μέσα. Ο συνάδελφος ε, κύριος ε, Ριβελίνη τοποθετήθηκε επί του θέματος. Έχουμε το non-paper της ε, Κομισιόν, το οποίο κατ' ουσίαν στο άρθρο 130 καθιστά σαφές ότι στα επιδοτούμενα δάνεια πρέπει να εφαρμόζονται τα χρηματοδοτικά μέσα τα επιδοτούμενα δάνεια θα ήθελα να ονομάζονται επιδοτούμενα δάνεια και όχι χρηματοδοτικά μέσα. Γιατί όταν λέμε χρηματοδοτικά μέσα, ο καθένα μπορεί να φανταστεί κάτι διαφορετικό. Μέχρι τώρα λοιπόν οι επιδοτήσεις των επιτοκίων κατ' ουσίαν ήταν επιδοτήσεις, καθαρές επιδοτήσεις. Και ε, ένα κράτος όταν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο κανονικά πρέπει να έρθει στην Κομισιόν και να το ανακοινώσει και να πάρει και άδεια. Η Κομισιόν λέει ότι εδώ θέλουμε να απλουστεύσουμε την όλη διαδικασία. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό, δηλαδή η Κομισιόν να αξιολογείται διαφορετικά από τα κράτη-μέλη. Και εμείς θα καταθέσουμε τροπολογία να υπάρχει ίση μεταχείριση. Στο άρθρο 131 ε, προβλέπονται πολλές ε, τροπολογίες για τα κριτήρια εισαγωγής ή αν θέλετε για, την, ε, για τον επιμερισμό των χρηματοδοτικών μέσων. Και όσον αφορά αυτό το χρηματοδοτικά μέσα, κανείς δεν το έχει ορίσει τι ακριβώς είναι και καλό θα ήταν να το ορίσει. Να λέμε ότι ξέρετε χρηματοδοτικό μέσο είναι το ΑΒΓ. Αυτή λοιπόν η έλλειψη ορισμού εμένα μου δημιουργεί πρόβλημα. Εγώ επιθυμώ διακαώ τον ορισμό και γιατί να μην υπάρχει ορισμός. Τα χρηματοδοτικά λοιπόν μέσα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές ε, της ε, διαφάνειας και της να μην υπάρχει έλλειψη αναλογικότητας. Αυτές είναι βασικά οι αρχές που διέπουν τα χρηματοδοτικά μέσα. Και πρέπει να σας πω ότι, πιστέψτε με, έχω αρκετή φαντασία για να Γνωρίζω ότι είναι τα χρηματοδοτικά μέσα. Αυτέ οι αρχέ λοιπόν που αναφέρονται, κατά την άποψή μου, δεν αρκούν. Προτείνονται λοιπόν νέε προποθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι η Ευρωπαϊκή Υπεραξία. Ε, Επίση, ε, το πλαίσιο ε, θα πρέπει να ισχύει εκεί όπου υπάρχουν διαφαινόμενοι κινδύνοι, να υπάρχει και η δυνατότητα της μόχλευσης και του πολλαπλασιασμού η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι φορεί πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Άρα δηλαδή, ε, όπως σας είπα, ε, το θέμα των χρηματοδοτικών μέσων και η διασύνδεσή τους με τα υπόλοιπα κονδύλια για μας είναι αποδεκτή. Η Κομισιόν, όπως σας είπα, επιθυμεί να έχει έναν ευρύ χαρακτηρισμό των χρηματοδοτικών μέσων, κάτι που όμως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει και δυστυχώς βρισκόμαστε και κάτω από πίεση χρόνου. Κατά τα άλλα ε, προσπαθούμε να ορίσουμε τον ε, ανώτατο ε, αποδεκτό κίνδυνο το αποδεκτό κίνδυνο σφάλματος. Επιθυμούμε να δημοσιεύονται οι διοικητικές διαπάνες και επιθυμούμε να έχουμε και ανταλλαγή απόψεων με τις καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές. Αυτό που είναι Παντελώ ασαφέ είναι τι θα κάνουμε ε, τα σημεία επαφής ε, που αφορούν τα χρηματοδοτικά μέσα και τα ΣΔΙΤ. Γιατί και τα ΣΔΙΤ ε, θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά μέσα. Για μένα λοιπόν αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί στα ΣΔΙΤ υπάρχουν πολλές και θεματικές εξελίξεις. Μέχρι τώρα λοιπόν είχαμε συμπράξει δημοσίου και δυτικού τομέα, ΣΔΙΤ, που ε, υπάγονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο όπου υπάρχει κανονισμός περί ε, προϋπολογισμού και όπου υπάρχει και κανονισμός περί προσωπικού. Τώρα όμως προτείνονται τρεις διαφορετικές μορφές ΣΔΙΤ. Ένα ΣΔΙΤ που θα αφορά άμεσα τι συνάψει έργου, το άρθρο 178, κατόπιν τα sui generis ε, που αφορούν ειδικέ περιπτώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ΣΔΙΤ που βασίζονται σε μια ειδική μορφή ιδιωτικού δικαίου του κράτους μέλους όπου μπορεί, κανείς, όπου μπορεί να συμμετέχει και μια εταιρεία. Άρα δηλαδή το θέμα είναι το εξή. Ε, στην Ισπανία, ας υποθέσουμε, ε, συστήνουμε μια εταιρεία περιορισμένη ευθύνη και εκεί εκπροσωπείται και η Κομισιόν ως μέτοχος. Αν θέλετε δηλαδή προκύπτει μία μορφή ε, κρατικού καπιταλισμού, μία μορφή που εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ μετά την ε, τόση του τείχους. Εγώ είχα θεωρήσει ότι ξεπεράσαμε αυτή τη φάση. Και μόνο αυτό, αλλά επανέρχεται και επανεθνικοποίηση της ε, ερευνητικής πολιτικής. Δηλαδή η Κομισιόν ως ευρωπαϊκό όργανο πηγαίνει στα κράτη-μέλη και μόνο αυτό αλλά υπάγεται και στο εθνικό, στο εκάστοτε εθνικό ισχύον δίκαιο. Και αυτό για μένα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εμείς λοιπόν είμαστε πρόθυμοι να εισάγουμε πολύ μεγάλες διευκολύνσεις για τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το μόνο ευρωπαϊκό ε, πρότυπο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή είναι όπως σας είπα sui generis ε, πρότυπο με νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι κανονισμό Συμβουλίου. Εμεί αυτόν τον κανονισμό του Συμβουλίου θέλουμε να τον εγκρίνουμε και στο μέλλον, αλλά με πάρα πολλέ διευκολύνσει που απομακρύνονται από την, ε, τον κανονισμό του ε, προσωπικού και τον κανονισμό περί προϋπολογισμού. Εκείνο όμως που δεν μου αρέσει είναι μια επανεθνικοποίηση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτόπου υπάγεται στο εκάστοτε ισπανικό, γερμανικό, ρουμανικό ή οποιοδήποτε άλλο δίκαιο και σε τελική ανάλυση, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι νομοθέτες, αν επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει να βάλουμε το ανώτερο όριο ε, και να μην δεχτούμε αυτή την επανεθνικοποίηση. Με λίγα λόγια λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα έχει ζητήσει το λόγο. Στρέφομαι και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα θέλατε το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης ή μήπως ήλθατε για να μας ακούσετε απλά. Ό,τι θέλετε. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο, ζητήστε τον και θα σας δώσω το λόγο. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους πρώτα. Έχουν μιλήσει ήδη δύο του ΕΛΚ, γι' αυτό θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Γκάιερ και μετά στην κυρία Ιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εισηγητές και τους δύο τους συναντέλφους Ριβελίνη και Γκρέσλε. Όλο αυτό το θέμα και τη διαδικασία εμείς ως σοσιαλδημοκράτες το παρακολουθούμε με συμπάθεια, με κατανόηση. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράσουμε και κάποιες δικές μας απόψεις που εν μέρει αφορούν τους εισηγητές και εν μέρει αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν αναφέρομαι στους εισηγητές. Κατανοώ πλήρως ότι είναι δύσκολο όταν τα κείμενα είναι ασαφή, ε, διότι όλη η διαδικασία ε, των συζητήσεων είναι ρευστή, προχωρά Είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς με αυτά τα δεδομένα σε κάποιο αποτέλεσμα. Έχοντας αυτά κατά νου, με το εξής. Το χρονοδιάγραμμα που ορίζετε εσείς, μήπως θα πρέπει να του βάλουμε δίπλα ένα μικρό ερωτηματικό. Τι σκοπεύετε να κάνετε με το χρονοδιάγραμμα. Προφανώς ε, δεν έχετε έτοιμη γνωμοδότηση της Κομισιόν και υποτίθεται παρόλα αυτά μέχρι τα τέλη του μήνα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγράφων. Έχω και μία ερώτηση περιεχομένου που αφορά στο θέμα της ε, διαπίστευσης. Ε, ίσως βέβαια ε, να μην τα έχω διαβάσει εκεί καλά. Κοιτάξτε, εξ όσων γνωρίζουμε έχουμε συστήματα διαχείρισης τα οποία τα έχουμε επιβάλει στα κράτη-μέλη και βέβαια αυτά ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη λειτουργικότητά τους και εφόσον εγκριθούν κατόπιν δείγματοληπτικά θα ερευνηθούν, θα εξεταστούν περαιτέρω από το ελεγκτικό συνέδριο και αφού γίνουν όλα αυτά μετά θα καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Αλλά αν θέλετε, ε, με τη δική μας τη γερμανική νοοτροπία αυτό σημαίνει διαπίστευση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως όμως εξελίσσεται η όλη συζήτηση, εγώ τελικά ε, καταλαβαίνω ότι μάλλον τα κρατη σκοπεύουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Και αν έχουν διαφορετικούς σκοπούς, παρακαλώ να μας τους πούν. Γιατί με το μέχρι τώρα ισχύον σύστημα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένο. Και τελικά, αν ε, τα κράτη-μέλη επιθυμούν κάτι άλλο, εγώ υποπτεύομαι, ξέρετε, αν το επιθυμούν, αυτό είναι λιγότερο έλεγχο. Θα με ενδιαφέρει, λοιπόν αυτή η, η άποψη Κομισιόν στο θέμα τη διαδικασία διαπίστευση. Και εγώ ως βουλευτής ε, ποια είναι τα πλεονεκτήματα που θα έπρεπε να διαβλέψω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ίσως το θέμα αυτό να έπαιξε ρόλο στο σεμινάριο που αναφέρατε και από το σεμινάριο και μετά είδα να εμφανίζονται πάρα πολύ εντυπωσιακοί όροι. Ακόμα και στην Επιτροπή Περιφερειών ε, ήρθα σε επαφή με όρους ε, που μου ήταν απόλυτα ε, καινούργοι ε, σε μένα που ασχολούμαι με θέματα προϋπολογισμού. Βεβαίως καταβάλλονται προσπάθειες να εξηγηθούν όλοι αυτοί οι όροι. Την προσπάθεια αυτή την κάνει η Επιτροπή, η Περιφερειακή Επιτροπή, αλλά ξέρετε κάπου τα πράγματα έχουν χαθεί, έχουν γίνει ένα καταλήξει σε χάος. Πανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της διαπίστευσης. Ποιες βελτιώσεις μπορεί να επιφέρει η διαπίστευση. Πρέπει να σας πω ότι τον ακούω από τα κράτη-μέλη ότι οποιαδήποτε μορφή κοινή διαχείρισης απορρίπτεται ε, ξέρετε συνάδελφοι, αυτό είναι τόσο προφανές όσο να λέμε ότι έξι τώρα είναι η μέρα και μετά αργότερα θα ανοιχτώσει. Πρέπει να, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τη Βόρεια Ορνανία Βεσφαλία. Εκεί θα ήταν κανείς ευτυχής αν καθίστατο δυνατό να εξευρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά κονδύλια να φτάσουν στον τελικό αποδέκτη χωρίς να χρειαστεί να υπάρξει επιπρόσθετη νομοθεσία. Γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, δημιουργούμε γραφειοκρατικό άχθος. Ο υπάλληλο πρέπει να κατανοήσει τους νέους νόμους και στη τελική ανάλυση δεν μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσον ε, τα νέα αυτά νομοθετήματα έχουν οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη χρήση. Ο υπάλληλο το μόνο που θα πει, α, καινούργια νομοθεσία, άρα αυτό είναι πολύ αρνητικό. Και επίσης ε, θέλω να σας πω ότι σχετικά με το σεμινάριο που αναφέρατε και με την επανεθνικοποίηση. Δεν ξέρω, πάνω σε αυτό δεν θέλω να τοποθετηθώ, αλλά θα ήταν ίσως σκόπιμο τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν περισσότερο με τις προτάσεις που κατατέθηκαν. Κατά τα άλλα, όσον αφορά το ε, αποδεκτό κίνδυνο σφάλματος, τον ανώτατο αποδεκτό κίνδυνο σφάλματος, θέλω να σας πω ότι εμείς ε, θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε λιγάκι το θέμα αυτό Βεβαίως ε, εδώ δεν μιλάμε για θρησκευτικό πόλεμο, κάτι άλλο. Ε, μιλάμε για ένα θέμα όπου θα καταλήξουμε κάπου, θα βρούμε κάποια λύση. Αυτά είχα να πω το παρόν και ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές και να τους ευχαριστήσω για αυτή την προσπάθεια τακτοποίησης αλλά και διαπίστωση για το που πάμε σε αυτή την αναθεώρηση του κανονισμού που επιφέρει νέες ευθύνες στο Κοινοβούλιο αλλά και ταυτόχρονα οδηγεί στην απλούστευση με την καλή της έννοια για να καταλήξουμε σε αυτήν τη νέα δομή του δημοσιονομικού κανονισμού να έχουμε λιγότερα λάθη. Και αυτό γιατί θα έχουμε λιγότερες ε, θα έχουμε λιγότερο, ε, λιγότερο μπερδεμένα πράγματα. Για το θέμα των ΠΠΠ και για το θέμα της ενιαίας θηρίδας ε, για αυτού του είδους της ενισχύσεις που οδηγούν ε, που θα αποτελούν ε, και πρόκληση για επενδύσεις στην έρευνα των ΜΜΕ, εγώ θα ήθελα να ξέρω αν με αυτή τη νέα διάταξη της ενιαίας θηρίδας δεν θα μπερδέψουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις ΜΜΕ οι οποίες ε, είχαν μία ειδική θηρίδα στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας. Αλλά αυτή τη στιγμή υποβληθεί αυτή η πρόταση η ΜΜΕ να μην χρειαστεί να εμπλακούν σε όλο αυτό το χάος που απαιτεί σήμερα η εκπόνηση ενός μεγάλου ερευνητικού σχεδίου. διότι κάποιος θα αισθανόταν πραγματικά ανήμπορος όταν μετά από την ενιαία θηρίδα που είχαν κερδίσει και κατακτήσει οι ΜΜΕ ξαναβρεθούνε σε μία φαραωνική διαδικασία που αφορά σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε πανεπιστήμια ή εργαστήρια. Τώρα, για τις εθνικές δηλώσεις. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτήν τη διαδικασία και πιστεύω ότι είναι καλή αυτή η συζήτηση που γίνεται, αλλά με, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια αυτές οι περίφημες δηλώσεις, εθνικές δηλώσεις οι οποίες χρησιμοποιούντουσαν ως πανάκια και λέγανε ότι ορίστε τα κράτη-μέλη θα μας δώσουν τα πάντα. Διαφάνεια και εγγύηση ότι το συγχρηματοδοτούμενο χρήμα βρισκόταν σε καλά χέρια. Σήμερα δεν πιστεύω ότι το πετύχαμε. Δηλαδή δεν πετύχαμε την απλούστευση αλλά ούτε και την επαλήθευση αυτού του μέσου. Διότι η πρακτική δείχνει και στις χώρες εκείνες που το ενέκριναν ότι ο Υπουργός ή οι Υπουργοί να υπογράφουν την απόφαση της ε, εκτέλεσης ε, της ε, δαπάνης, αυτό για μας δεν είναι εγγύηση για μας ότι τα χρήματα ξοδεύτηκαν σωστά και είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις πέρυσι. Πρέπει να δούμε λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε από κοινού με την Επιτροπή να βρούμε ένα σύστημα τεχνολογικό. Πετύχαμε αυτό να λειτουργεί το σύστημα για τις ατομικές ενισχύσεις στη Γεωργία και θα έπρεπε οι διάφοροι πρωταγωνιστές σε τοπικό, επαρχιακό, περιφερειακό επίπεδο θα έπρεπε λοιπόν όλοι αυτοί να είναι καταγεγραμμένοι και να έχουμε εμείς μία μηχανογραφημένη εικόνα για το ποιος χρηματοδοτείται, πώς ξοδεύει το χρήμα χωρίς να μπερδεύουμε ακόμη περισσότερο τις περίφημες εθνικές δηλώσεις. Ρωτώ την Κομισιόν αν έχει καμιά ιδέα χωρίς να υπερφορτώνουμε άλλα επίπεδα και να μην περιμένουμε εμείς ο κάθε δήμαρχος, ε, αντιδήμαρχος της Άνω Μαγούλας να υπογράφει ένα χαρτί και να λέει ορίστε διαχειριστήκαμε τα χρήματα σωστά και εμείς να το πιστεύουμε. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να έχουμε ένα μηχανισμό για να ξέρουμε πώς χρησιμοποιείται το κοινοτικό χρήμα. Και για τα νέα δημοσιονομικά μέσα εγώ συμφωνώ με αυτό το νέο Ταμείο Εγγύησεων, με τις διευρυμένες ε, αρμοδιότητες της ΕΤΕ. Συμφωνώ ότι όλα αυτά μας θέτουν μπροστά σε νέες ανάγκες, δηλαδή με ευρωπαϊκές αποφάσεις. όπου δημιουργούνται νέοι όροι για τον κοινοτικό αλλά και για τον εθνικό προϋπολογισμό. Χρειάζεται λοιπόν και εμείς να έχουμε κάποιες νέες μεθόδους, νέα μέτρα για να μπορούμε να κρίνουμε. Διότι εμείς έχουμε όλα αυτά τα κατεπήγοντα μέτρα λόγω της κρίσης αλλά δεν έχουμε τις εγγύησεις προς τον πολίτη για να εγγυθούμε ότι είναι αποτελεσματική η χρήση των κονδυλίων και ότι ελέγχουμε αυτά τα κονδύλια. Πρέπει να δούμε αν μπορούμε και εδώ να φανταστούμε κάτι ούτω ώστε το ελεγκτικό συνέδριο, εθνικό ή ευρωπαϊκό, να μπορεί να ελέγχει αυτά τα μέσα. διότι εμείς αποφασίσαμε ένα σωρό νέα δημιουργικά και φάνταστα μέτρα αλλά δεν έχουμε φανταστεί τον αντίστοιχο έλεγχο αυτών των μέτρων. Λοιπόν, θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Δεν φαίνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω λίγο να αντισωμαδοποιήσω ομαδοποιήσω θέμα και να δώσω ίσως κάποιες πρώτες απαντήσεις όχι απαντώντας στους ίδιους τους βουλευτές, αλλά στα θέματα τα οποία, σχολιάζοντας τα θέματα τα οποία έθεσαν τώρα. Το θέμα των μέσων, των χρηματοδοτικών μέσων, το θέμα της συνέργειας ιδιωτικού δημόσιου τομέα, η κοινή από κοινού διαχείριση, οι εθνικές δηλώσεις, το θέμα της πιστοποίησης και το θέμα του ανεκτού λάθους, επίπεδου, ανεκτού επίπεδου λάθους, όπως επίσης και της μονοαπευθυντικής θηρίδας. Γενικά ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε στη διάρκεια μιας φάσης επεξηγηματικής. Οι προτάσεις τις οποίες κάνουμε είναι σε στάδιο ανάλυσης και παρουσίασης. Οι αναλύσεις αυτές, το είπε άλλωστε η εισηγήτρια, περνούν μέσα από μία έγγραφα, από non-paper και προς τα δύο σκέλη τα δημοσιονομικά, τα υπεύθυνα της αρχής της υπεύθυνη για τον προϋπολογισμό. Για να ξεκινήσω από τα πιο απλά θα έλεγα. Ανεκτά επίπεδα κινδύνου. Όλο και περισσότερο είναι σαφές ότι η πρόταση η οποία περιλαμβάνεται στον δημοσιονομικό κανονισμό, στην πρόταση δημοσιονομικού κανονισμού δεν είναι αποδεκτή για το νομοθετικό κομμάτι και θα πρέπει η έννοια αυτή να περάσει σε μια διαφορετική αρχιτεκτονική ενός διαχειριστικού πλέον μέσου. Η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών λοιπόν της Επιτροπής θα κάνει προτάσεις πρώτα στους μεμονωμένους επιτρόπους και στη συνέχεια στο σύνολο των επιτρόπων έτσι ώστε να χαρακτηριστεί πλέον η διαδικασία αυτή μέσω διαχείριση στο δημοσιονομικό κανονισμό στα πλαίσια των κατεξουσιοδότηση διατακτών, δηλαδή των γενικών διευθυντών. Αυτοί είναι οι διατάκτες κατεξουσιοδότηση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακούσαμε λοιπόν το μήνυμά σας και θα το μεταφέρουμε σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι εκεί δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Σχετικά τώρα με την εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η κυρία Κρέσλα σωστά παρατήρησε ότι προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το μοναδικό υπάρχον πρότυπο, το οποίο είναι ένα πρότυπο που εφαρμόζεται και στις πρωτοβουλίες κοινή τεχνολογίας, οι οποίες θα πρέπει να, υπόκονται, να υπόκεινται συγγνώμη, και στον κανονισμό και στο ε, ε, δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό οδηγεί αυτά τα GDI σε, μία θα έλεγα πάρα πολύ δύσκολη εκκίνηση λειτουργίας. Ακούσατε και εσείς τους εκπροσώπους αυτών των GDIs οι οποίοι διαμαρτύρονται ε, για το μακρόσυρτο των διαδικασιών εκκίνησης. Και όμως οι δράσεις αυτές είναι σημαντικότατες για την ευρωπαϊκή έρευνα. Πήραμε επίσης μέρος σε πολλές συναντήσεις με τους διευθυντές αυτών των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλειών και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς προτιμούν Γι' αυτό άλλωστε και προτείναμε δύο διαφορετικά άλλα μοντέλα, δύο διαφορετικά πρότυπα. Το λεγόμενο sui generis, Το sui generis είναι ένας οργανισμός ο οποίος θα δημιουργηθεί μετά από κοινοτικέ αποφάσεις. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε εν μέρη να μην υπόκειται στον κανονισμό και αυτό θα ικανοποιήσει φυσικά τους υπεύθυνους των GDIs γιατί ξέρουμε ότι αν θέλουν ας πούμε ένα συμπληρωματικό πρόσωπο πρέπει να περάσουν από κάποιες διαδικασίες βαρύτατες και περιπλοκότατες. Κάτι το οποίο τους παρεμποδίζει στη σωστή τους εργασία. Το θέμα είναι να υπάρξει μια κοινοτική απόφαση η οποία να δημιουργεί αυτές τις εταιρικές σχέσεις δημόσιος ιδιωτικός τομέας. Ταυτόχρονα όμως να επιβληθεί στους συγκεκριμένους οργανισμούς μια σειρά δημοσιονομικών ρυθμίσεων η οποία θα αποτελεί την σωστή εγγύηση για την χρηστή οικονομική διαχείριση των GDIs. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ζητηθεί από τον κόσμο της έρευνας εδώ και πολύ καιρό. Και αυτό είναι κάτι που θα επιτρέψει αυτές οι κοινέ πρωτοβουλίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα προτείνουμε επίσης και SDIC, PPP, στα οποία να εκφεύγουν του ιδιωτικού δικαίου, ανάλογα με το πού θα εγκαθίστανται βέβαια. Στην ουσία, Υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο ξέρω καλά, το οποίο λειτουργεί σήμερα. Κατανοώ βέβαια ότι μπορεί κάποιος να έχει επιφυλάξει σε σχέση με αυτή τη μορφή λειτουργίας των ΣΔΙΚ. Ίσως να προσπαθήσω να εξηγήσω κάπως περισσότερο στην ε, κυρία Γκρέσλε συγγνώμη, και στον κύριο Ριβελίνη τον τρόπο που λειτουργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση το συγκεκριμένο ΣΔΙΚ. Είναι ένα περιορισμένο θα έλεγα παράδειγμα αλλά παρόλα αυτά κατανοώ ότι μπορεί να υπάρχουν επιφυλάξεις. Λοιπόν, για τα PPP, στα ΣΔΙΚ, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει ουσιαστικά τεθεί από τους ίδιους τους εκπροσώπους του ερευνητικού κόσμου Έχουμε λοιπόν την πρόθεση με κάθε τρόπο να διευκολύνουμε τη δημιουργία αυτών των PPPs. Ανάμεσα στα τρία πρότυπα υπάρχει ένα εν λειτουργία, ένα το οποίο είναι κοινοτικού χαρακτήρα και το οποίο θα λειτουργήσει και ένα τρίτο για το οποίο υπάρχει ανάγκη περισσότερων εξηγήσεων. Γρήγορα τώρα για τη μοναπευθυντική θηρίδα έτσι όπως περιλαμβάνεται στο έγγραφο εργασίας των εισηγητών. Η συγκεκριμένη αυτή θηρίδα εμπνέεται θα έλεγα άμεσα των προτάσεων που έγιναν πέρυσι και στις αρχές της φετινής χρονιάς για το πλαίσιο της έρευνας. Δεν πρόκειται για μια περίπτωση υποχρεών, υποχρέωσης μάλλον αυτών οι οποίοι χρηματοδοτούνται να περνούν μέσα από μια τέτοια θηρίδα. Απλά Πρόκειται για, μια, για ένα επίπεδο ερμηνείας των εγγράφων, ενιαίας όμως μορφής ερμηνείας για όλες τις γενικές διευθύνσεις που ασχολούνται με την έρευνα, γιατί διαπιστώσαμε ότι ανάλογα με τη γενική διεύθυνση προς την οποία απευθύνονται οι ερευνητές, αντιμετωπίζουν μερικές φορές διαφορετικού τύπου ερμηνείας των δημοσιονομικών κανονισμών, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι η μοναπευθυντική θηρίδα είναι μια λύση η οποία θα ελεγχθεί τους επόμενους μήνες και ελπίζω να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Συμφωνώ με την κυρία Γιάλα Σέντερ ότι μια τέτοια θηρίδα για όλους τους τομείς παρέμβασης του προϋπολογισμού του γενικού στην έρευνα είναι κάτι το πολύ ε, φιλόδοξο, περίπλοκο και φαραωνικό όπως λέει ο μιλητής. το να υπάρξει το λεγόμενο clearance committee, τη μια προαδιοδοτική επιτροπή, ε, ίσως ε, κάτι τέτοιο να μπορέσει να βοηθήσει κάπως καλύτερα αυτούς οι οποίοι καλούνται να επωφεληθούν των προβλέψεων του Γενικού Προϋπολογισμού στο μέλλον. Τώρα έρχομαι στα ε, οικονομικά μέσα, στα χρηματοδοτικά συγγνώμη μέσα. Εδώ η Επιτροπή είναι αλήθεια ότι υπερέβαλε στο λιτό της παρουσίασης των προτάσεών της. Και μάλιστα και στον προηγούμενο δημοσιονομικό κανονισμό ήμασταν ακόμα πιο ξηροί και λιγότερο επεξηγηματικοί. Και απλά δεν είχαμε ε, προβλέψει τις εξαιρέσεις, τις επιδοτήσεις που προβλέφθηκαν εκ των υστέρων. Πρέπει λοιπόν αυτές τις εξαιρέσεις να τις ε, αφαιρέσουμε από το κεφάλαιο των ε, επιδοτήσεων και να τους δώσουμε ένα διαφορετικό καθεστώς. Γιατί όπως είπαν ορισμένοι από εσά, όπως θεωρούν ορισμένοι από εσά, οι δημοσιονομικές και οι οικονομικές γενικότερες συνθήκες που σοβούν σήμερα οδηγούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά όλο και περισσότερο. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη εδώ να διευκρινιστούν κάποια πράγματα καλύτερα και να συντονίσουμε τα βιολιά μας και εμείς ε, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Πράγματι, όπως είπε η κυρία Γκρέσλε, θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα αυτά τα οικονομικά μέσα που χρησιμοποιούμε θα κάνουμε λοιπόν κάποιες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, προς, τις, τους δύο κλάδους, ε, το, τους δημοσιονομικούς, για να δώσουμε τις απαιτούμενες εξηγήσει. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να επαναλάβουμε αυτά τα οποία προϋπήρχαν στον προηγούμενο δημοσιονομικό κανονισμό, πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 130 του προηγούμενου κανονισμού. Θέλουμε να ορίσουμε καλύτερα ποια είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν. Ε, σαν παράδειγμα ε, εκπτώσεις στα δάνεια, στο κόστος των επιτοκίων, όπως επίσης και στα μέσα χαμηλού κινδύνου. Καθορίζουμε δηλαδή καλύτερα το τι ε, περιλαμβάνεται στο άρθρο 130 και το οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στον δημοσιονομικό κανονισμό και στην κατεξουσιοδότηση δευτερεύουσα πράξη από την οποία θα προέλθει ο κανονισμός λειτουργίας. Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε επίσης και τις συνθήκες μέσω των οποίων προσφεύγουμε σε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις δηλαδή. Η κυρία Γκρέσλε αναφέρθηκε σε κάποιες από τις προϋποθέσεις αυτές, απαριθμό κάποιες από αυτές, Υπάρχει άλλωστε και ένα έγγραφο το οποίο έχει αποσταλεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τον έλεγχο όλων αυτών των προτάσεων. Θα πρέπει λοιπόν τα χρηματοδοτικά μέσα να προσφέρουν μια κάποια αξία επιπλέον στην κοινοτική δράση να χρήζουν βελτιώσεως οι προτάσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν, να μην δημιουργούνται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, να λειτουργούν κινητοποιώντας τις ερευνητικές δυνατότητες μέσω των δυνατοτήτων του κοινοτικού προϋπολογισμού. Εδώ πολλαπλασιαστή μπορεί να είναι από 2 μέχρι 20 θα πρέπει επίσης η οντότητα προς την οποία επιβεβαιούμε ή εκχωρούμε αν θέλετε τη διαχείριση αυτής της ε, δημοσιονομικής διαχείρισης να έχει τους ίδιους στόχους και τα ίδια συμφέροντα με τους ε, στόχους και τα συμφέροντα τα οποία εκφράζει η κοινοτική πολιτική μέσω της οποίας χρηματοδοτείται. Και η το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να επιβεβαιεί κάθε φορά εάν οι στόχοι αυτοί ε, στηρίζονται και εξυπηρετούνται από τους κανονισμούς. Τώρα για την απόσβεση αυτών των ε, δανείων και τα λοιπά, για μια κάποια χρονική περίοδο υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα. Ε, κάποια από τα χρήματα αυτά τα οποία δεν χρηματοποιούνται κάποιοι ζητούν να μην επιστρέφουν στο γενικό προϋπολογισμό ή να μην καταλήγουν απευθεία στα ταμεία τα εθνικά. Και υπάρχει επίσης και μια ολόκληρη σειρά άλλων προϋποθέσεων, οι πιο σημαντικές από αυτές είναι να μην τίθενται θέματα απλά έκπληνσης χρημάτων. Θα πρέπει οι χρηματοδοτήσεις αυτές να χρησιμοποιούνται για στόχους μη τρομοκρατικούς, να εξελίσσονται οι δράσεις αυτές σύμφωνα με τις φορολογικές συνθήκες οι οποίες σε κάθε περίπτωση ισχύουν Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που θα έχουμε με τις χρηματοδοτούμενες οντότητες. Ταυτόχρονα, λάβαμε το μήνυμά σας και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σωστή ενημέρωσή σας για το τι συμβαίνει με όλα αυτά. Επιθυμούμε πράγματι να προβλέψουμε σε μια έκθεση η οποία είναι ισχνή προς το παρόν αν και υπάρχει μια ετήσια έκθεση η οποία να αναφέρεται στις δραστηριότητες αυτών των οργανισμών, στις επιδόσεις των οικονομικών μέσων, των χρηματοδοτικών μέσων, στο τι επιστρέφει στα χρηματοδοτικά μέσα μέσω των επιστροφών, στο ποιος είναι ο πραγματικός παλαπλασιαστικός συντελεστής, μια ετήσια έκθεση εν πάση περιπτώσει η οποία θα δημοσιεύεται κατά τα μέσα του μηνός Ιουνίου μάλλον προς τις και θα δίδεται στις νομοθετικές αρχές. Λοιπόν, αυτά για τα χρηματοδοτικά μέσα. Νομίζω ότι πράγματι κάνουμε μία κάποια προσπάθεια να καλύψουμε τις επιθυμίες της κυρίας Γκρέσλε για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να οξύνουμε τα μέσα παρέμβασής μας, αλλά παρατηρώ με ικανοποίηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στρέφεται θετικά, διάκειται εν πάση περιπτώσει θετικά, εφόσον αναγνωρίζεται βέβαια και ο ρόλος του και καθορίζεται σωστά ο συγκεκριμένος ρόλος. Ένα τελευταίο σημείο, η κοινή διαχείριση. Η κυρία Γκρέσλερ Για μια μισή μέρα πήρε μέρος ή παραβρέθηκε αν θέλετε και πήρε μέρος όσο μπορούσε εν πάση περιπτώσει στο σεμινάριο για την κοινή διαχείριση. Και την ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Νομίζω ότι η κυρία Γκρέσλε κατάλαβε ποιες είναι οι δυσκολίες των κρατών μελών και εδώ δίδω απαντήσεις και προς τον κύριο Γκάιερ σχετικά με το τι προβλήματα έχουν τα κράτη-μέλη με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αποκοινού διαχείριση τι είναι. Τα γεωργικά ταμεία, τα διαρθρωτικά ταμεία, η αλληλεία, που ανήκει βέβαια στα γεωργικά, και κάποια άλλα επιμέρους μέσα σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής. Τι. Προσπαθούμε να βρούμε λοιπόν κοινέ δομές διαχείρισης και γι' αυτό κάνουμε προτάσεις οι οποίες προσωμιάζουν με το πρότυπο που χρησιμοποιείται στο γεωργικό τομέα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στα κράτη-μέλη. Γιατί τα κράτη-μέλη έχουν δομές, ιδιαίτερα για τα διαφορετικά ταμεία, οι οποίες είναι λειτουργικές. Και το ξεκαθαρίζω αυτό. το ότι υπάρχει μια διαχειριστική υπηρεσία, το ότι υπάρχει μια υπηρεσία πιστοποιητική και υπάρχει και μια υπηρεσία εκ των υστέρων ελεγκτική. Τα κράτη-μέλη λοιπόν μας είπαν ότι ο πιστοποιητικός οργανισμός πριν φτάσει άμεσα η πρόταση και η, διάταξη, η διαταγή πληρωμής, το διατακτικό πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι χρήσιμο για να μειωθεί το ποσοστό λάθος. Εμείς λοιπόν κατανοήσαμε τα κράτη-μέλη και προσπαθήσαμε στο μέτρο του δυνατού να προτείνουμε μέσω του συνόλου των επιτρόπων αυτό που είναι αποδεκτό από τα κράτη-μέλη να μην θίξουμε ιδιαίτερα τις υπάρχουσες εν λειτουργία δομές. Η πιστοποίηση τώρα. Εδώ, εδώ είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα πρόσφατο, υπάρχει στις τομεακές πράξεις και διαχωρίζει από τη μία τα διαφορετικά και από τα γεωργικά. Η διαδικασία πιστοποίησης έχει σαν στόχο τον έλεγχο του οργανισμού στο οποίο εμπιστευόμεθα τα κοινοτικά χρήματα έτσι ώστε ο οργανισμός αυτός να είναι απολύτως σε θέση να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στα διαφορετικά ταμεία αυτό το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα γεωργικά ταμεία το κράτος μέλος αναλαμβάνει την εγγύηση της πιστοποίησης και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο Α, ο Β, ο Γ οργανισμός είναι σε θέση να διαχειριστεί σωστά το κοινοτικό χρήμα. Αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε έχει μεικτό χαρακτήρα, δηλαδή κοινή διαχείριση σημαίνει και κοινή ευθύνη στον καθορισμό των οργανισμών οι οποίοι θα τύχουν ε, τις επιλογής αυτής. Θέλουμε δηλαδή τα κράτη-μέλη να εμπλακούν περισσότερο στον ε, ορισμό αυτών των διαφορετικών μηχανισμών διαχείρισης του κοινοτικού χρήματος και θέλουμε επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εγκαταλείψει όλα αυτά στα χέρια των κρατών μελών και να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία πιστοποίησης και αυτή. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με κάτι το οποίο προσωπικά θεωρώ όταν παρουσιάστηκε στα πλαίσια των συμπειρασμάτων του σεμιναρίου προκάλεσε κάποιες θετικές αντιδράσεις από πλευράς των κρατών μελών γιατί εκεί υπήρχαν και ελεγκτές και διαχειριστές εκπρόσωποι των κρατών μελών. Αυτό το οποίο είναι το πιο δύσκολο στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας είναι να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της διαδικασίας που ξεκινά από αυτούς οι οποίοι δίδουν τα χρήματα και ε, καταλήγει στην ε, έκδοση αν θέλετε της πιστοποίησης που δίνει η αρμόδια υπηρεσία. Γι' αυτό ακριβώς καταλήγουμε και στις λεγόμενες δηλώσεις αξιοπιστίας των διαχειριστών. Μπορούμε να τις ε, αναφέρουμε αυτές τις ανακοινώσεις και σαν δηλώσεις διαχείρισης αν θέλετε αλλά αυτό που έχει σημασία είναι οι διαβεβαιώσεις οι οποίες μας δίδονται και προέρχονται από τους κατατόπους διαχειριστές για να κατατίθενται σε μία περίοδο η οποία να είναι χρήσιμη στους γενικούς διευθυντές. Οι διευθυντές παρουσιάζουν την γενική έκθεση δραστηριότητά τους στο τέλος του μηνός Μαρτίου και αμέσως μετά εκείνη η διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στην απαλλαγή. Συνεπώς θα πρέπει αυτά τα οποία λαμβάνουμε, οι πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε από τους κατατόπους διαχειριστές, να συμπίπτουν χρονικά ή να καλύπτουν χρονικά την περίοδο ε, ε, ε, για την οποία δίδει τις διαβεβαιώσεις που του ζητούνται ο Γενικός Διευθυντής. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να μετακινήσουμε την περίοδο για την οποία παίρνουμε τις διαβεβαιώσεις αυτές από πλευρά των κρατών μελών προς την κατεύθυνση κάλυψης ε, του οικονομικού έτους που προηγείται Τη έκθεση δραστηριοτήτων των Γενικών Διευθυντών. Και εδώ έχουμε πρόβλημα χρονισμού, έχουμε πρόβλημα πρακτικών ε, δημοσιονομικού ελέγχου που οργανώνονται από τους διαχειριστές αλλά και από τους ελεγκτές εκ των υστέρων. Υπάρχει ένα πρόβλημα χρονισμού, δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά θα πρέπει να έχουμε αρκετά στοιχεία στη διάθεσή μας, έτσι ώστε η δειγματοληψία η οποία εκτελείται από τους έλεγκτες ε, να είναι αρκετά ευρεία για να δίνει σωστά αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε με κάτι το οποίο σε μία πρώτη φάση μας οδήγησε στην πρόταση που έχουμε μπροστά μας έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα την 1η Φεβρουαρίου ή έστω τις 15 Φεβρουαρίου για να έχουν οι γενικοί διευθυντές ένα μήνα σύντομο μήνα για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν τα στοιχεία αυτά στη γενική έκθεση δραστηριοτήτων τους. Το πρόβλημα αυτό το υπογράμμισε και η κυρία Γκρέσλε και ο κύριος Βιβελίνη. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις γύρω από αυτό στα πλαίσια του σεμιναρίου. Προσπαθήσαμε εμείς να πάμε λίγο προς τα πίσω την ημερομηνία που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία αυτά έτσι ώστε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να αναλάβει τα στοιχεία αυτά ε, να τα διαχειριστεί και να τα παρουσιάσει πριν από την τελική έκθεση 15 Ιουνίου. Κατανοήσαμε λοιπόν ότι για αυτήν την αποκοινού διαχείριση θα πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν. και εδώ θα σας κάνουμε κάποιες προτάσεις, θα κάνουμε κάποιες προτάσεις και στην πολιτική αρχή του Συλλόγου των Επιτρόπων, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και των κρατών μελών και τις δικές σας παρατηρήσεις που ακούσαμε. Το πρόβλημα είναι εδώ να μην μείνουμε με το παρόν σύστημα συνολικά ως έχει, γιατί υπάρχουν πολύ συχνά ποσοστά λάθος τα οποία είναι πάρα πολύ υψηλά. Όχι η έκθεση φέτος, αλλά τις άλλες χρονιές η έκθεση για το 2009 τα δείχνει όλα αυτά. Στο παρελθόν τα ποσοστά λάθους βέβαια ήταν πολύ ψηλότερα από ό,τι η τελευταία έκθεση. Αυτά σας εξήγησα λοιπόν ότι είδαμε τι θέλουν τα κράτη-μέλη, ήταν παρούσα και η κυρία Γκρέσλε, οι αντιδράσεις τους ήταν πάρα πολύ αρνητικές, δεν θέλουν να αλλάξουν τις πρακτικές τους, πρόκειται αν θέλετε για ένα ρεφλεξ κατανοητό, αλλά το οποίο δεν ικανοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό θα επανέλθουμε. Λυπάμαι γιατί μίλησα πάρα πολύ. Όχι τόσο, αλλά αλλά παρόλα αυτά ήταν νομίζω χρήσιμο για να κατανοήσουν οι παρόντες ευρωβουλευτές ποιο είναι το περιεχόμενο των προτάσεών μας. Eh, eh, Είναι πολύ θετικό το ότι απαντήσατε αναλυτικά στις ερωτήσεις των διαφόρων συναδέλφων και αυτό και γιατί είχαμε χρόνο και γιατί ήταν χρήσιμο. Και σας ευχαριστώ προκαταβολικά αν μπορέσετε να έρθετε σε επαφή με τους εισηγητές για να συζητήσετε συγκεκριμένα πράγματα θα χρειαστούν ακόμη μερικοί μήνες ε, για να ολοκληρωθούν ε, οι εργασίες. Ο κύριος Μπόρστοκ από το Ελεγχητικό Συνέδριο. Πρόεδρε, ε, δύο πολύ σύντομα μήνυματα από τον πιστό σας φίλο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το πρώτο μήνυμα. Το δικαστήριο γνωμοδότησε για αυτή την πρόταση και αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε, με τα χαρά θα το κάνουμε. Δεύτερο μήνυμα. Η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει κάποιες ε, τροποποιήσεις ε, ως προς τον εξωτερικό έλεγχο. Δηλαδή αυτά που εμείς κάνουμε και όπως μπορείτε να δείτε στη γνωμοδότησή μας ορισμένες εξ αυτών των προτάσεων ε, τις ε, χαρακτηρίζουμε κακές και άλλες πάλι κάκιστες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι τόσο ο κύριος Ριβελίνη όσο και η κυρία Γκρέσλε και η δική σας επιτροπή και η Επιτροπή Προπολογισμών θα λάβει υπόψη τις ε, τις προτάσεις μας και νομίζω ότι είναι προς το όφελος της Ευρώπης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δουλεύει αποτελεσματικά και φαντάζομαι ότι η δική σας Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γι' αυτό ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε ελπίζω να μην μακρηγόρησα Αν θέλετε να το στείλετε να βάλετε το μήνυμα σε, σε ένα μπουκάλι θα πετάξουμε το μπουκάλι στον ωκεανό Κυρία Γκρέσλερ, κύριος Ριβελίνη. Κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μα είπατε. Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί κανεί να το ακούει όρου ολοκλήρω, αλλά ούτε για 10 λεπτά δεν μιλάει το ε, ελεγκτικό συνέδριο. Τι κρίμα. Ελπίζω, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, να βρούμε και κάποιες λύσεις. Αλλά ας μην αυταπατώμεθα. Τις λύσεις που δεν θα βρούμε τώρα, δεν θα τις έχουμε καν μέχρι το 2020. Γι' αυτό λοιπόν ανησυχώ με αυτά που είπε ο κύριος Κάιρ. Κοιτάξτε κύριε Κάιρ, εμείς θέλουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, αλλά αν τελικά εσείς μας κατακλείσετε με τροπολογίες, προφανώς αυτό θα δυσχεράνε τη δουλειά μας. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια μεγάλη μεταρρύθμιση με πάρα πολλά και νέα σημεία. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ε, θέλω όμω να σα πω ότι σε τελική ανάλυση ούτε και εμεί δεν είμαστε ικανοποιητικά προετοιμασμένοι για αυτή τη μεταρρύθμιση. Α πούμε, τα περίφημα GTIs που αναφέρθηκαν και προηγουμένω. Γι' αυτό ζήτησα το λόγο. Τα GTIs έκαναν την αξιολόγηση αλλά και πάνω σε μια βάση δεδομένων που δεν αρκεί. Και αυτό το λέει η αξιολόγηση. Λέει, διαβάσαμε την έκθεση Σάρμπα ε, και την άλλη έκθεση για τις joint undertakings ε, στα Clean Sky ή στο πρόγραμμα Artemis. Δύο δηλαδή. Ε, εγώ διάβασα και τις δύο αυτές εκθέσεις και κατόπιν τούτου θεωρώ ότι εδώ, εκεί μάλλον, πρόκειται για ένα ευχολόγιο, το οποίο ευχολόγιο έχει προσκρούσει σε δίκο ε, αότα. Τώρα, με εκπλήσει αυτό, αλλά από την άλλη δεν πρέπει κανείς ε, να με κατηγορήσει ότι και εγώ δεν έχω κατανόηση για την ερευνητική κοινότητα. Όμως δεν είναι σωστό όλα αυτά τα θέματα να τα υιοθετήσουμε. Νομίζω αυτό ακολουθεί λάθος κατεύθυνση. Γιατί σε τελική ανάλυση εμείς θα είμαστε χαμένοι. Εμείς θα χάσουμε τον έλεγχο. Όλα αυτά τα πρότυπα που υπάρχουν στον ερευνητικό τομέα, μα ποιος θα τα ελέγχει. Εμείς θα υποστούμε τις συνέπειες ε, και ε, επειδή έχουμε αναπτύξει ορισμένες ε, τεχνικές, ε, δεν θέλουμε να τις ε, απορρίψουμε. Επειδή λοιπόν και εγώ θέλω να εξοικονομώ τις δυνάμεις μου, επιμένω να διατηρήσουμε τη θέση μας και νομίζω ότι τελικά όλοι θα παραμείνουν ικανοποιημένοι. Ως έχει το θέμα τώρα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αφήσουμε. Και να δείξω και ένα άλλο θέμα που έδειξε και ο συνάδελφος κυρίως Ριβελίνη το θέμα των κατεξουδότηση πράξεων. Δεν θα δώσουμε μια γενική εξοδότηση, λευκή επιταγή για τις εφαρμοστικές διατάξεις τώρα. Με τις συνθήκες της Λισαβόνας τα πράγματα έχουν αλλάξει και η Κομισιόν πρέπει να μας δει που ακριβώς χρειάζεται περαιτέρω κατεξουσιοδότηση πράξης. Και μας ανέφερε 100 άρθρα όπου πιστεύει ε, ότι χρειάζεται περαιτέρω νομοθετικό έργο. Ε, πολλά αυτά τα 100 άρθρα. Θα το εξετάσουμε λοιπόν, θα δούμε κατά πόσο πράγματι ε, χρειάζονται 100 ή λιγότερα. 60 προτείνει η Κομισιόν όπου επιθυμεί οι εφαρμοστικές διατάξεις που ήδη υπάρχουν να συμπεριληφθούν στον ε, δημοσιονομικό κανονισμό. Ε, θέλω να δείξετε κάποια κατανόηση. Ε, δεν πρόκειται για μικροδιαχείριση, αλλά πρόκειται για μια νομική κατάσταση που έχει τροποποιηθεί. Μιλάμε για ε, το δικαίωμα της συναπόφασης, το χρονοδιάγραμμα. Κοιτάξτε, αυτή η Επιτροπή επηρεάζεται τα μάλα από την απαλλαγή. Κύριε Μπόστοκ, όσο θαραλέοι και αν είμαστε, τελικά το μόνο που μπορέσαμε να κερδίσουμε είναι ένας μήνας. Δύο μήνες από την Κομισιόν, δύο από το ελεγκτικό συνέδριο, τέσσερις από εμά και κερδίσαμε, εμείς προτείνουμε λοιπόν η απαλλαγή από την Ολομέλεια του Απριλίου, μάλλον από την Ολομέλεια του Μαΐου να πάει στην Ολομέλεια του Απριλίου, λέει η κυρία Κρέσλε. Γιατί επιθυμούσαμε να πάμε πιο κοντά στο Δεκέμβρη και επιθυμούσαμε να πούμε ε, το έτος νη συν ένα επιθυμούσαμε να έχουμε κλείσει. Τώρα πάντως σας λέω ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμως ότι είναι σημαντικό να ε, περιορίσουμε λιγάκι τη διαδικασία που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα έχουμε ίσως μια περισσότερη ε, συνεδρίαση γιατί θα πρέπει να επιταχύνουμε λιγάκι. Εμείς λοιπόν σας λέω ε, παρετούμεθα από τέσσερις εβδομάδες ή άλλοι από δύο εβδομάδες ο έκαστος. Όμως σας παρακαλώ να μην αρχίσετε το να μαγειρεύετε το χρονοδιάγραμμα είτε θα το κάνουμε αυτό που σας είπα είτε όχι γιατί όλα αυτά είναι συνάρτηση και πολλών άλλων ημερομηνιών. Άρα όλα μαζί ή τίποτα και ε, επιθυμώ τα αποτελέσματα τη απαλλαγή να χρησιμοποιηθούν και στον προπολογισμό. Γι' αυτό επιθυμώ να υπάρχει περιορισμό ε, του χρονοδιαγράμματο. Εγώ νομίζω ότι οι καλέ ιδέε επιβραβεύονται και αυτό που κάνουμε ω διαδικασία ποτέ δεν έχει ξαναγίνει. Δεν είναι η πρώτη ανάγνωση όπου κάτι στέλνει το Συμβούλιο, κάτι στέλνει η Κομισιόν, κάτι θέλουμε εμεί. Οι καλέ ιδέε επιβραβεύονται και είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτε γιατί πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία. Ε, και για πρώτη φορά ε, προβλέπουμε τα κατα τα πιστευματικά ταμεία. Αυτά είναι επιθυμία του Κοινοβουλίου, ακριβώς όπως και η μόνο απευθυντική θηρίδα για την ερευνητική κοινότητα. Η Κομισιόν, ε, το ότι επανέρχεται τώρα, αυτό το βρίσκουμε σωστό και αυτό είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός ε, όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Όσον αφορά όμως τα καταπιστευματικά ταμεία, εμείς επιθυμούμε να ε, περιοριστούμε στην κοινή διαχείριση και μετά από το 2020 και εφεξής ε, μπορούμε ίσως αν θέλετε να εφαρμόζουμε ε, περισσότερο αυτή τη δυνατότητα που μας προσφέρεται. Ευχαριστώ ο εισηγητής. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συντομεύουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε όμως να, κάνουμε διαστικές δουλειές. Υπάρχουν πολύ σημαντικά σημεία, το ανέφερε και η συνάδελφος ε, Γκρέσλερ, οι εντεταλμένες πράξεις, οι θέσεις ορισμένων θεσμών, θεσμικών οργάνων, θα επιταχύνουμε όσο μπορούμε, θα ανασκομποθούμε, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Περιμένουμε εμείς τα SMS του ελεγκτικού συνεδρίου. Λοιπόν, ας μας στείλει αυτά τα μηνύματάκια και εμείς θα τα λάβουμε υπόψη. Είμαστε έτοιμοι με την κυρία Γκρέσλερ να συναντήσουμε και την Επιτροπή. Θα ανακουσκουμποθούμε, θα σκεφτούμε. Το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κλείνουμε με το σημείο 27. Έχουμε ένα διαδικαστικό της κυρίας Αγιάλα, η οποία ζήτησε, πολύ σύντομα την παρακαλώ, να κάνει ορισμένες παρατηρήσεις για το σημείο 33 της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στον Γενικό Προϋπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΟΚΕ. Η κυρία Γιάλα θέλει μια προφορική τροπολογία σχετικά που να εξηγεί γιατί δεν θέλει να, να δώσει αυτή τη στιγμή την απαλλαγή στην ΟΚΕ. Παρακαλώ να ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο συντομότατα, διότι μετά έχουμε στις 5.30 τη συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Δεν μπορούμε να χάνουμε ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την αναφορά διότι διότι εγώ ήθελα και ζήτησα από τον εισηγητή να αναβάλουμε την απαλλαγή του Γενικού Προϋπολογισμού για την ΟΚΕ και αυτό γιατί στις 11 Μαρτίου η Όλαφ ξεκίνησε μία διαδικασία παραβίασης κατόπιν ε, καταγγελιών για κακή διαχείριση και ανομαλίες στην ΟΚΕ. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι παρκώς σοβαρά για να τα λάβει η υπόψη της ε, η Επιτροπή μας. Εγώ παρουσίασα ένα κείμενο στα αγγλικά για την τροπολογία 2 στην έκθεση Ριβελίνη όπου προσπαθώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για τα προβλήματα στην ΟΚΕ. και που τον Απρίλιο του 2009 είχαν οδηγήσει σε διάφορες ε, παρατυπίες και είχαν οδηγήσει επίσης ένα από τα μέλη της ε, ΟΚΕ να υποβάλει μια καταγγελία στην ΟΛΑΦ και η ΟΛΑΦ να ξεκινήσει μια διαδικασία. Εγώ θα έλεγα να το αναβάλουμε και αν η Όλαφ μας πει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τότε εμείς ε, να ψηφίσουμε. Αλλά πρώτα ας μας ενημερώσει η Όλαφ, διότι άμα εκκρεμεί διαδικασία δεν ε, νομίζω ότι είναι λογικό εμείς ε, να εγκρίνουμε. Από όσα τώρα εγώ έχω διαβάσει στο φάκελο και από όσα γνωρίζω, Υπάρχουν ε, προβλήματα στην ΟΚΕ. τα οποία ξεκίνησαν από τον Απρίλιο του 2009 και όχι τον Δεκέμβριο του 2009, όπου είχε ξεκινήσει μία πειθαρχική διαδικασία και εκ διαπιστώθηκαν ε, ατασταλίες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ζητάω για να αποφύγουμε τέτοια πράγματα αναβολή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς ε, να κάνει καμιά παρατήρηση. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν διμερείς ε, ε, Έρχεται πίσω ο κύριος Ριβελίνη να τον περιμένουμε, επανέρχεται και ο κύριος Σόντεργατ ήθελε και αυτός να υποβάλει μια πρόταση, καμιά ερώτηση. Εγώ παρουσίασα αυτές τις προτάσεις για να τις λάβετε υπόψη σας. Ο κύριος Ριβελίνη, τι έχετε να πείτε για την πρόταση της κυρίας Αγιάλα. Είναι πρόβλημα για σας. Εγώ δεν συμφωνώ γιατί στις 11 Μαρτίου όντως ξεκίνησε μια διαδικασία της Όλαφ μετά από καταγγελίες ενός πρώην ε, υπαλλήλου Ισπανού του Μόσες Μπένγκάρτεν. Όλοι θέλουμε να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι ευθύνε, αλλά η απαλλαγή η άρνηση της απαλλαγής, η, συγγνώμη, η αναβολή της απαλλαγής θα δημιουργούσε κολλήματα στην Όλαφ αντί να τη διευκολύνει. Και η αναβολή της απαλλαγής ε, νομίζω ότι θα ήταν κάτι το, ε, το οποίο θα ενίσχυε από τη μια μεριά την ερευνητική διαδικασία. Αλλά από την άλλη μεριά όμως υπάρχει περίπτωση η Όλαφ να κλείσει τον έλεγχο και να αρχιοθετήσει την υπόθεση. Εμείς μετά μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να κρίνουμε τις αποφάσεις της Όλαφ, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένη αυτή η πρόταση. Εγώ πιστεύω, λέει ο Πρόεδρος, ότι δεν πρέπει να μακρηγορούμε. Η κατάσταση είναι σαφής. Λοιπόν, αύριο ψηφίζουμε. Σημείο 33, οκ. Μία από τις ε, πρώτες ε, ψηφοφορίες είναι αν δίνουμε ή όχι την απαλλαγή. Και η πλειοψηφία θα αποφασίσει αν θα δώσουμε απαλλαγή ή όχι. Αν υπάρχει πλειοψηφία αύριο για να αναβάλουμε την απαλλαγή, τότε η κυρία Γιάλα που το ζητάει θα παρουσιάσει μία προφορική ε, ερώτηση θα το αιτιολογήσει και μετά θα δούμε αν η προφορική τροπολογία της κυρίας Αγιάλα μείνει ή όχι. Λοιπόν, το πρώτο είναι η απαλλαγή ή όχι. Τελειώσαμε με την δημόσια συνεδρίαση. Σταματάει το web streaming και ξεκινάει η συνεδρίαση και, των, και κλεισμένων των θερών. Όποιο είναι άσχετο με τη συνεδρίαση παρακαλώ να βγει. Eh,